Ελήφθησαν κάποιε αποφάσει από του συντονιστέ στις τελευταίες Δεν είχαμε συνεδριάσει επιτροπή μετά τις συνεδρίες των συντονιστών. Να σε ενημερώσω 16 Δεκεμβρίου συνεδρίες των συντονιστέ Ελήφθησαν αποφάσει. Η Ντανούτα Χίμπνερ είναι η συγγήτρια για την έκθεση για τη Οργανική Συμφωνία για καλύτερη θέσπιση νομοθεσία. Αποφασίσαμε σε αυτή τη συνεδρίαση ότι η αποστολή στην Αθήνα τη ΑΦΚΟ θα γίνει 30 Μαρτίου Απριλίου. 30-31 Μαρτίου και 1 Απριλίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά τις συστάσεις αυτές θεωρούνται εγκεκριμένες και θα ανακοινωθούν οι συστάσεις σήμερα της σημερινής συνεδρίας των συντονιστών ελήφθησαν αποφάσεις σήμερα. Πρώτα απ' όλα, έκθεση ΑΦΚΟ για την ερμηνεία και εφαρμογή της Ιοργανικής Συμφωνίας για καλύτερη θέσπιση νομοθεσίας. Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε συνεργασία ΑΦΚΟ με τη Ζούρη σύμφωνα με το άρθρο 55 αν ζητήσει η Τζούρη κάτι τέτοιο και οι σοσιαλιστές θα είναι υπεύθυνοι για την έκθεση και με στέντες Μπέσο πρότεινε τον Ρίτσαρτ Κόρμπερτ σαν εισηγητή από πλευρά ΣΑΦΚΟ αποφασίσαμε και για τη γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 54 με την Επιτροπή Προπληγισμού και ΚΟΝ για το δημοσιονομικό δυναμικό της Ευρωζώνης η γνωμοδότηση πάει στο ΕΛΚ θα διορίσουν εισηγητή και λήφθηκε απόφαση να ετοιμάσουμε γνωμοδότηση, η Επιτροπή μας να ετοιμάσει γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 53 για έκθεση προπολογισμού για την πολιτική συμμετοχή του Κοινοβουλίου για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και οι σοσιαλιστές θα διορίσουν εισηγητή. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών λοιπόν θα ετοιμάσει τη σχετική έκθεση. Και κάτι άλλο να σας πω. Θα ήταν λογικότερο να το λέγαμε το πρωί. Το πρωί όμως είχαμε συνάντηση με την Προεδρία. Εν τω μεταξύ συναντήθηκα και τον Πίτερ Γκιουγέρ, τον πρέσβη της Ολλανδίας, αρχές Ιανουαρίου συζητήσαμε θέματα που ανέφερε και ο ε, Υπουργός για το δικαίωμα εξέτασης. Τους ενημέρωσα λοιπόν για τις εκθέσεις Μπρέσο, Μπροκ, Βερχόφστατ και Γκίγκουλτ και Ραμόν για την ηλεκτρονική δημοκρατία να ξέρει η Προεδρία τι κάνουμε. Γιατί θα υπάρχουν και επαφές και θα εμπλακούν στις προσπάθειες και για τον εκλογικό νόμο ενημέρωση των προσβευτή, ποια είναι η προσέγγιση μας, τι περιμένουμε από την Προεδρία. Συζητήσαμε και το θέμα της Οργανικής Συμφωνίας για καλύτερη νομοθεσία. Συζητήσαμε την επικείμενη συνάντηση της ΚΟΖΑΚ επί Ολλανδικής Προεδρίας θα διεξαχθεί στη Χάγη η συνάντηση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Συμμετέχω και εγώ λόγω της θέσης μου Συζητήσαμε αυτά τα θέματα λοιπόν με τον κύριο Προσβευτή. Αυτά. Περιμένουμε την άφηξη του Υπουργού. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, εκτός αν έχετε κάτι εσείς να πείτε. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Καμιά άλλη πληροφορία. So we wait for Minister Schmidt. Περιμένουμε τον Υπουργό Νίκολας Σμιτ. What item 11? Σημείο 11, πού είναι το σημείο 11? Uh, ah, Α, απαλλαγή. Δεν είναι εδώ ο αρμόδιος. Το 12 το κάναμε. Τα διάφορα, δεν έχω διάφορα. Άρα τα καταφέρνουμε. 14 είναι η επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 του μηνός. Πώς το ξέρουμε αυτό. Α. Λοιπόν, ξεμπερδέψαμε με αυτά. Δεν χρειάζεται να τα εξετάσουμε μετά. Τελευταίο σημείο για σήμερα θα είναι το 11 της ημερήσιας διατάξης.

Συνάδελφοι, είναι πέμπτη απόγευμα και μεταδίδεται διαδικτύου ευτυχώ η συνεδρίαση. Όσοι δεν είναι παρόντες μπορούν να ακούσουν. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Εκτιμούμε το ότι ήρθε ο υπουργό Νίκολας Σμιτ μετά την ολοκλήρωση της ε, Λουξεμβουργιανής Προεδρίας να μας πει τις απόψεις του. Να μας πει πώς βλέπει την Ευρώπη σήμερα από την σκοπιά του. Είπε ότι θα αισθάνεται ελεύθερος άνθρωπος. Να δούμε πώς μηνά ένας ελεύθερος άνθρωπος στους ευρωβουλευτές. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς, σας ευχαριστώ που με καλέσατε μετά την Προεδρία. Μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να επανέρχομαι εδώ σε εσά και να αισθάνομαι, πώς να πω, σαν να μην έχουν τελειώσει όλα. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να πω, αισθάνομαι και μια κάποια ανακούφιση. Το ευχαριστήθηκα να είμαι παρόν στο Κοινοβούλιο και μόνο στη δική Επιτροπή και σε άλλες επιτροπές συμπεριλαμβανομένης της Ολομελίας. Ναι, και στη συνάντηση με εθνικά κοινοβούλια, ναι, ναι, ναι, ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Δεν θέλω να μακρηγορήσω όσον αφορά τη Λουξεμβουριανή Προεδρία. Ήταν μια περίοδος ε, γεμάτη από δραστηριότητες, τραγωδίες, μεγάλες προκλήσεις που και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όπως είπαν και κάποιοι, Ίσως ποτέ δεν έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν τόσες πολλές απειλές και τόσα πολλά ερωτηματικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετανάστευση και η κρίση για τη μετανάστευση είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε. Και με τους συναδέλφους από την Ολλανδία οι συνάδελφοι από την Ολλανδία θα πρέπει να συνεχίσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν σταματάει και το πράγμα. Ε, τώρα συζητάμε ουσιαστικά και θεμελιώδη στοιχεία τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται με το Σέγγεν, που είναι βασικό στοιχείο τη ευρωπαϊκή οικοδόμηση και τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τι γίνεται με την αλληλεγγύη εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτή η έννοια, αν σημαίνει κάτι ακόμα. Δέχτηκε επιθέσεις αυτή η αλληλεγγύη και δεν βρήκαμε ακόμα τις σωστές απαντήσεις για τους πρόσφυγες, αλλά όχι μόνο εκεί. Αντιμετωπίσαμε και άλλες προκλήσεις. Και οι ελεύθερες και δημοκρατικές κοινωνίες μας δέχονται προκλήσεις. Καταρχάς, από όλες αυτές τις απειλές, λόγω τρομοκρατίας, αυτό που ζήσαμε στις αρχές της ε, χρονιάς, της περασμένης χρονιάς και στο τέλος της, ήταν ε, δραματικό. Αμφισβητεί τις ελεύθερες και ανοιχτές κοινωνίες μας. Και όμως υπάρχουν επίσης και μελά, μερικά μεγάλα ερωτηματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις ελεύθερες και ανοιχτές κοινωνίες. Και όμως εκεί δράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι από τις θεμελιώδεις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές. Που δεν, είναι, δεν θα ήθελα να πω ότι έχει αμφισβητηθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τουλάχιστον έχουν ε, πει κάποια ερωτηματικά σε κάποιες, από κάποιες χώρες. Και βεβαίως ε, ερωτήσεις είναι δύσκολε αυτές και απαντήσεις θα πρέπει να δώσει και το Κοινοβούλιο. Τι γίνεται με τις βασικές ελευθερίες, τι γίνεται με τα βασικά δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα ελευθερία του τύπου, τα ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τέτοιου τύπου ερωτηματικά που είναι θεμελιώδη. Όχι μόνο στα κράτη-μέλη τη Ένωση, αλλά για την ίδια τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέκυψαν όλα αυτά τα ερωτήματα και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε εμείς. Θα πρέπει οι επόμενες προεδρίες να ασχοληθούν. Εμείς προσπαθήσαμε να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Το πρώτο είναι η διαθεσμική συμφωνία. Εκεί τουλάχιστον καταφέραμε να σημειώσουμε μια επιτυχία, να κλείσουμε αυτό το ντοσχέ. Κάναμε μια διαπραγμάτευση και μια ολοκλήρωση, επιτυχή αυτής της νέας διαθεσμικής συμφωνίας. Το έχετε συζητήσει? Όχι, θα το συζητήσετε εν συνεχεία. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες τότε για αυτό το σημείο, γιατί το έχει κάνει ο διαπραγματευτής σας. Θέλω καταρχήν όμως να ευχαριστήσω και το Κοινοβούλιο και το διαπραγματευτή του για την πολύ θετική και επικοδομητική στάση τους και τη συμμετοχή τους στη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Φερχόφσταντ. Χάρη στη θέση που πήρε, χάρη στην ε, θετική του στάση και απόψεις, καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία. υπάρχουν και κάποια σημαντικά θέματα που μας απασχόλησαν εμάς ως Προεδρία, που ενδιαφέρουν φυσικά και το Συμβούλιο, ή τουλάχιστον μια ευρύτατη πλειοψηφία κρατών στο Συμβούλιο. Δεν ήταν το Λουξεμβούργο εκεί, αλλά η Προεδρία που εκπροσωπούσε το Συμβούλιο, που ήταν ο διαπραγματευτή. Και ποια, ποια είναι αυτά τα σημεία. Πρώτον, να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων να μην έχουν ε, αντιπαλότητες μεταξύ τους και για να λειτουργεί σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε ένα καλό σύστημα εργασίας και συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Και αυτή η νέα διαθεσμική συμφωνία νομίζω ότι αποτελεί καλή βάση για κάτι τέτοιο. Θέλουμε όμως επίσης να εξασφαλίσουμε ότι οι αρμοδιότητες που εγγυάται η συνθήκη ή οι συνθήκες δεν θα μπορούσαν έμεσα να περιοριστούν ή να αμφισβητηθούν μέσω μια τέτοια συμφωνίας. Όλοι θέλουμε καλύτερη νομοθεσία, καλύτερε ρυθμίσει, θέλουμε μια απρόσκοπτα λειτουργούσα Ένωση αποτελεσματική, μη γραφειοκρατική, που δεν διαθετεί νομοθεσία που κανένα δεν θέλει και δεν χρειάζεται. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Γι' αυτό όμως. Και αυτή η συμφωνία την εξασφαλίζει αυτή την ισορροπία. Εξασφαλίζει μια καλύτερη, πιο αποτελεσματική λειτουργία. Αποφεύγουμε νομοθετήματα άχρηστα ή το να βάζουμε σε νομοθετήματα στοιχεία που δεν χρειαζόμαστε. Απ' την άλλη όμως, εμείς θεωρούσαμε ότι είναι σαφές ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τι σημαίνει η απουσία της Ευρώπης, το κόστος της μη Ευρώπης. Όπως το λέμε. Και διαπιστώσαμε σε πολλούς τομείς ότι το κόστος αυτός είναι πολύ ψηλότερο από το να έχουμε υπερβολικά επαχθή νομοθεσία. Όταν δεν υπάρχει Ευρώπη, υπάρχουν 28 διαφορετικές νομοθεσίες. Υπάρχει σύγχυση για την εσωτερική αγορά. Υπάρχει έλλειψη εναρμόνισης κτλ. λοιπά Και αυτό κοστίζει και για τις επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο αυτό που συχνά αναφέρεται ότι η Ευρώπη κοστίζει και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Δεν θέλω να πω ότι δεν συμβαίνει ποτέ. Μπορεί να συμβεί μερικές φορές. Αλλά η απουσία της Ευρώπης, μιας καλής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μιας καλύτερης εναρμόνισης μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών και των εθνικών αγορών, μερικές φορές αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θέλαμε να επαναφέρουμε στο πνεύμα αυτής της συμφωνίας και τελικά καταφέραμε μία συμφωνία που είναι και ισορροπημένη και θα βοηθήσει σε μία πιο λειτουργική Ευρώπη και σε πιο εύρυθμα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Δύο λόγια για ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ καλύτερη διακυβέρνηση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια. Έχετε ετοιμάσει και μια έκθεση για τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του δυναμικού της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Και έχουμε την ευκαιρία να το... Είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε στην ανταλλαγή απόψε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θυμάζετε ή τουλάχιστον συζητάτε την προετοιμασία μιας έκθεσης για να ενσωματώσουμε την διακυβερνητική συμφωνία για τη σταθερότητα, συντονισμό και την διακυβέρνηση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εδώ το θέμα μιας καλύτερη και πιο στεναρή διακυβέρνηση κυρίως στην Ευρωζώνη και στην καρδιά της Ευρωζώνης. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για μένα, όχι μόνο ω υπουργό υπεύθυνο για ευρωπαϊκέ υποθέσει, αλλά και υπουργό για κοινωνικέ υποθέσει. Οπότε διαβάζω και το είπατε και σε κάποιου λόγου, και εσεί κυρία ότι θα πρέπει να σκεφτούμε αν αυτή η συνθήκη είναι αρκετή. Και μήπω είναι μονόπαντη. Γιατί α, εστιάζει μόνο στην καλύτερη διακυβέρνηση. Σε μία πτυχή τη μάλιστα. Δεν λαμβάνει υπόψη άλλε. Και εγώ θα βάζα και την κοινωνική διάσταση εδώ. Και γι' αυτό προσπάθησα να το κάνω και άκουσα κάποια κράτη-μέλη να λένε να μου αποδίδουν προθέσεις που δεν τις είχα. Ότι βάλτε την... Ε, θέλουμε να έχουμε συναντήσεις των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωζώνης. Αλλά νομίζω ότι κάπου πρέπει να βάλουμε και αυτό το στοιχείο, ε, το κοινωνικό δηλαδή, ε, στο better governance. Και τώρα πάμε σε κάτι άλλο. τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Κάναμε μια ανταλλαγή απόψεων γι' αυτό. Έγινε μια άτυπη ανταλλαγή στα πλαίσια του Κορεπέρ και οι δύο συνεισηγητές συμμετείχαν στο Κορεπέρ. Ήταν ένα πρόγευμα εργασίας όπου οι δύο συγητέ του Κοινοβουλίου συναντήθηκαν με το Κορεπέρ. Τώρα υπάρχει η δική σας έκθεση επιτάπητο και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εκεί πέρα. Το θέμα πια δεν είναι το Λουξεμβούργο από μόνο του. Εγώ εξακολουθώ να σας υποστηρίζω, αλλά αυτό που προτείνει αυτή η έκθεση είναι σαφέστατη βελτίωση για τις ευρωπαϊκές εκλογές αλλά είναι βελτίωση, γιατί δίνει και μεγαλύτερη νομιμότητα σε αυτές τις εκλογές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε και το συζητήσαμε αυτό στο παρελθόν με το Γιώργο Λάινεν, το πώς δηλαδή θα, ψη... θα πείσουμε τον κόσμο να ψηφίσει, το πώς θα τον πείσουμε ότι έχει σημασία η ψήφος του και έχει σημασία να ψηφίσει αυτές τις εκλογές. Νομίζω ότι με τις μεταρρυθμίσεις που προτείνεται οι οποίε είναι πολύ σημαντικέ, θα πρέπει να περάσουν, το πετυχάνουμε σε κάποιο βαθμό. Αλλά ξέρετε ότι είναι μια ειδική διαδικασία και μάλιστα πολύ περίπλοκη. Βασιστείτε όμω πάνω μα στην υποστήριξή μα για αυτό το θέμα. Το τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι η Εκταστική Επιτροπή. Ομολογώ ότι εδώ δεν προχωρήσαμε όσο θα θέλαμε. Προσπαθήσαμε να επανεκκινήσουμε τη συζήτηση. Είχαμε μια καλή συζήτηση με τον εισηγητή. Κάναμε και κάποιες ανταλλαγές μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Και ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και φαντάζομαι ότι θα συμβουλεύσετε του διαδόχους μας στην Ολλανδική Προεδρία να συνεχίσει τι εργασίε από αυτού. Εμείς νομίζω ότι δώσαμε νέα πνοή στο θέμα αυτό. Καλό είναι να αρχίσουμε την εργασία από αυτού και να βρούμε τα κοινά σημεία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ε, Γιατί θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Σας ενθαρρύνω και σας υποστηρίζω και για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ας αρχίσουμε τώρα την ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Σέφλιν πρώτος, μετά η κυρία Μπρέσο, μετά ο κύριο Γιολάινεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και εσά, κύριε Υπουργέ που προσήλθατε πάλι ενώπιον μας ε, σήμερα και με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τις απόψει σα. Το Λουξεμβούργο έχει προεδρεύσει κάτι επανάληψη. Κάθε νέα προεδρία ωστόσο συνεισφέρει και κάτι καινούριο. Έχετε δίκιο που λέτε ότι πρόκειται από τις πιο δύσκολες περιόδους που έχει περάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια μικρή ερώτηση και μια δεύτερη μεγαλύτερη, ίσως να μην απαντήσετε στη δεύτερη. Η πρώτη είναι για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, που νομίζω ότι είναι ακόμα στα Σπάργανα. Μιλήσαμε για αυτήν σήμερα το πρωί με την Ολλανδική Προεδρία. Πώς την βλέπετε εσείς. Εξακολουθώ να λαμβάνω το λεγόμενο feedback από τα κάτω, από μη κρατικές οργανώσεις, από πολίτες και από τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι ακόμη. Το άλλο ερώτημα που ίσως να μην θέλετε να απαντήσετε είναι για την αλληλεγγύη και αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποίησατε και εσείς. Εμένα μου φαίνεται ότι η αλληλεγγύη θα λειτουργήσει μόνο, θα υλοποιηθεί μόνο, εάν αποτελέσει την έκβαση μιας συζητήσεως. Δεν μπορεί να επιβληθεί η αλληλεγγύη. Αυτό που έγινε φέτος σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης έγινε αντιληπτό ως ένα δικτάτ. Γι' αυτό και υπάρχει αντίσταση που ε, εν μέρει μάλιστα σημειώθηκε στη διάρκεια της Λουξεμβουργικής Προεδρίας. Διερωτώ με άλλο, άραγε πώς την αισθανθήκατε εσείς αυτήν την ε, συγκεκριμένη περίοδο. Η πρόεδρος Χιούπνερ, η Μερσέντε πρώτα. Ευχαριστώ στο όνομα της ομάδας των σοσιαλιστών, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τη Λουξεμβουργική Προεδρία βεβαίως για τις εργασίες της Είχαμε πολλές ευκαιρίες να συζητήσουμε μαζί σου για σημαντικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως πάντα ε, εκτιμήσαμε πολύ τις δεσμεύσεις, την στάθευσή σου για τα θεσμικά θέματα για μια καλύτερη Ευρώπη καθώς και για τα κοινωνικά θέματα. Μεταξύ άλλων, χάρη και στις προσπάθειες της δικές αλλά και όλων, κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε την διαθεσμική συμφωνία και από αυτή τώρα θα εργαστούμε ως κοινοβούλιο για να την περάσουμε στις δραστηριότητες μας. Δύο θέματα τώρα για τα οποία θα ήθελα να ερωτήσω και να ζητήσω τη γνώμη σου. Πρώτο, μας μίλησες για μια ομάδα εργασίας που εγκύπτει στο θέμα της βελτίωσης των σχέσεων με τις εθνικές βουλές. Για την πράσινη κάρτα. Αυτή η ομάδα εργασίας έχει καταλήξει σε συμπεράσματα, έχει ολοκληρώσει το έργο της θα συνεχίσει και υπό άλλε προεδρίες. Είχαμε κάποιες ειδήσει, αλλά πολύ περιορισμένες. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω εάν πρόκειται να γίνει κάποια πρόταση. Δεύτερο, εφιστώ την προσοχή της ε, Λουξεμβουργική κυβέρνησης, όχι πια της Προεδρίας, για ένα θέμα καλύτερης οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης και κυρίως στις κοινωνικές πτυχές. Κάνουμε κατά βάση δύο προτάσεις με τον Έλμαρ Μπρόκ στην έκθεση που θα συζητήσουμε πολύ σύντομα. Αφενός θα ζητήσουμε από την Κομισιόν να φτιάξει ένα σύνολο κριτηρίων για την αξιολόγηση της απόδοσης των προσπαθειών των χωρών μελών για τα κοινωνικά θέματα και εκεί το πάλι ποια είναι η γνώμη σου και το δεύτερο θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα πραγματικό κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο να ξεκινήσει να επαναφέρει τη συζήτηση ότι η Ευρώπη είναι μια κοινωνική οικονομία και όχι μόνο των αγορών θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν τη γνώμη σου και ως ε, Υπουργό Εργασίας. Γνωρίζω ότι αυτά τα θέματα σας απασχόλησαν στην Προεδρία. Να απαντήσετε. Για την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Εγώ την υποστηρίζω την ιδέα αυτή. Ήμουν και μέλος στην συνέλευση τότε και θεωρώ ότι είναι σημαντικό στοιχείο και μάλιστα θα πρέπει να γίνει πιο σημαντικό ακόμη για να επιτρέψει προσέγγιση των πολιτών στην Ευρώπη και να τους δώσει και κάποια δυνατότητα άσκηση επιρροή σε ευρωπαϊκέ πολιτικές. Δυστυχώ ακόμη δεν έχει φτάσει στο επίπεδο αυτό. Αυτό είναι ατυχές. Νομίζω ότι πρέπει να επανεξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας της πώς μπορεί να εφαρμοστεί λοιπόν, πώς μπορεί να τη εσύ, Εμεί θα το στηρίξουμε αυτό. Χρειάζεται να εξυγχρονιστούμε και χρειάζεται να επανεπινοήσουμε τα δημοκρατικά μα συστήματα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο μάλιστα. Να μην αγνοούμε ότι υπάρχει ένα κενό, μια απόσταση ανάμεσα στους πολίτες και στους θεσμούς. Χωρίς να περιορίζομαι μόνο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το ίδιο χάσμα υπάρχει και με τους εθνικούς θεσμούς. μπορούμε να φτιάξουμε έτσι μια πιο συμμετοχική δημοκρατία. Και αυτό ήταν και το νόημα της πρωτοβουλία εκείνης. Να δοθεί δηλαδή στους Ευρωπαίους πολίτες το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους, τις επιθυμίες τους και να εξηγούν σε ποια πράγματα αποδίδουν σημασία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έτσι λαμβάνονται και αποφάσεις. Αλλά πάντως η ιδέα ήταν να δοθεί όθηση αυτή, σε αυτό το project δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Νομίζω ότι υπάρχει μια μελέτη που έγινε. Αναμένουμε τώρα να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ε, επιτρέπω σε αυτόν να συστήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν πρόκειται για κανένα περιορισμό του δικαιώματός τους του μονοπωλίου της πρωτοβουλίας. Χρειάζεται να προσαρμόσουμε και λίγο τη λειτουργία της Ένωσης από τη σκοπιά αυτή. Είμαι λοιπόν απολύτως υπέρ. Η Κομισιόν τώρα να έρθει να κάνει προτάσεις και στη βάση των προτάσεων που έχουν εκπονηθεί. Ασφαλώς βέβαια θα χρειαστεί να συζητήσουμε το θέμα αυτό και στο Συμβούλιο, διότι είναι σαφές ότι στο Συμβούλιο θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια δεύτερη δημοκρατική όθηση και η πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο συνεισφορά. Για τη δεύτερη ερώτησή σου θα είναι σύντομο. Σύμφωνο ότι η αλληλεγγύη δεν είναι κατά κάποιο τρόπο νομικό εργαλείο. Η αλληλεγγύη θα πρέπει πρωτίστως να είναι ένα πριν ε, στα γαλλικά, να έρχεται από τα μέσα δηλαδή. Θα πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν και δρούν οι χώρες μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες εξ αυτών. Η αλληλική λοιπόν είναι μια βασική αρχή λειτουργίας της Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι σε τι αναφέρεστε Εννοείται την ε, έννοια αυτή των ποσοστώσεων, που δεν μου αρέσει τόσο πολύ ω έννοια, αλλά αυτό εννοείται. Καμιά φορά χρειάζεται να οργανωθεί η ελληνική πράγματι. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια στάση τέτοια από όλους μας. Θα αρκεστώ σε αυτά, αλλά συμφωνώ ότι δεν γίνεται αυτό μόνο με εφαρμογή κανόνων. Χρειάζεται ένα συνολικότερο πνεύμα που να κατησχύσει στην Ένωση. Και αυτό το πνεύμα είτε χάνεται είτε γίνεται πιο χαλαρό. Όταν συμβαίνει αυτό νομίζω ότι μπαίνουμε σε δύσκολα νερά. Αυτό νομίζω ότι γίνεται τώρα μάλιστα. Τώρα για τις εθνικές βουλές. Τέτοια έκθεση δεν υπάρχει τουλάχιστον όποιον του Συμβουλίου. Μπορεί να κυκλοφορεί μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων. Δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να παίξουν ένα ρόλο, σημαντικό μάλιστα. Υπάρχουν προβλέψεις στη συνθήκη που τους αποδίδουν αυτόν τον ρόλο. Και αυτό που είπα στην συνάντηση με τις εθνικές βουλές είναι το εξή. Δεν μπορούν να αποτελέσουν νέο ευρωπαϊκό θεσμό. Γιατί τέτοιο ενδεχόμενο θα ανατρέψει τις ισορροπίες ε, που ενυπάρχουν στο σύστημα. <clears throat> Νομίζω δώσαμε στις Εθνικές Βουλές πολλά νέα δικαιώματα, καλώς πράξαμε και εγώ είμαι ανοιχτός στη σκέψη ιδιαίτερα για την Ευρωζώνη, πώς μπορούν να συμμετάσχουν περισσότερο τα Εθνικά Κοινοβούλια με κατάθεση ιδεών και αυτό ίσως είναι σημαντικό εκεί Τώρα όμως το να δώσουμε στα εθνικά κοινοβούλια ή σε ένα εθνικό κοινοβούλιο, σε ορισμένα εθνικά κοινοβούλια, ένα δικαίωμα άρνηση κυρίας, αυτό όπως είπα θα ανατρέψει την ισορροπία του συστήματος. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και γνωρίζεις καλά τι εννοώ, Mercedes. Σε ό,τι αφορά τώρα την διακυβέρνηση, governance, το είπα και πριν, ότι όντως πρέπει να την βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση. και να την καταστήσουμε περισσότερο δημοκρατική. Νομίζω ότι η διακυβέρνηση στερείται δημοκρατικότητας και πράγματι εκεί στην Ευρωζώνη υπάρχει ρόλος για τα, για τα εθνικά κοινοβουλία. Το πώς μπορεί να γίνει ή πώς να, μπορεί να εκφραστεί, δεν θέλω τώρα να προβάλλω ιδέες, αλλά όντως υπάρχει ανάγκη να εμπλακούν τα εθνικά κοινοβουλία, διότι η οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση υπησέρχεται και στους εθνικούς προϋπολογισμούς και επομένω στο πεδίο κυριαρχίας των εθνικών κοινοβουλίων. Άρα πρέπει να συμμετάσχουν και αυτά και βεβαίως και μεγαλύτερη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τα κοινωνικά τώρα κριτήρια η θέση μου είναι ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε μια ισορροπία. Όταν έχουμε προπολογισμού, δημοσιονομικές πολιτικές, μακροοικονομικές πολιτικές, Όλα αυτά έχουν μεγάλες επιπτώσεις στα κοινωνικά μας συστήματα, στα συστήματα κοινωνικής ευημερίας. Δεν μπορούμε να πούμε αυτά είναι ξεχωριστά τώρα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αυτό ε, επιφέρει μια αντίφαση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η κοινωνική διάσταση λοιπόν πρέπει να εγκαθιδευτεί και να οριστεί σαφέστερα. Και η ιδέα να υπάρξει ένα είδος πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων έχει ενδιαφέρον. Διάβασα και άκουσα τα όσα είπε η Επιτροπή, η Κομισιόν δηλαδή, και ο Πρόεδρος της. Όμως ήδη κυκλοφορούν πολλές δηλώσεις και διακηρύξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1989, διάβασα μάλιστα σχετικά ένα άρθρο, το 1989 εγκρίθηκε, η υποκαλική Προεδρία τότε, ο χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων. Έχουμε και χάρτε και διακηρύξει, πολλά τέτοια πράγματα. Όταν μιλούμε για κοινωνικά δικαιώματα, ο λόγο μα θα πρέπει να είναι σοβαρό και νομικά δεσμευτικό. Οι δεμοί είναι ωραία λόγια όλα αυτά, αλλά δεν αλλάζουν τίποτε. Αυτή είναι, αυτός είναι, αυτή είναι η πραγματική συζήτηση. Και έρχομαι εδώ σε αυτό που είπε, το κοινωνικό πρωτόκολλο ή κοινωνικό συμβόλαιο. Όταν μιλούμε και μάλιστα για να εντάξουμε την διακυβερνητική συνθήκη μέσα σε ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συζητήσουμε και κάποιο είδου ε, συνθήκη ή πρωτόκολλο ή πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων όπως θέλετε πέστε το και με την ευκαιρία αυτή θα διεξαχθεί η συζήτηση αν απλά περιοριστούμε σε μια διακήρυξη ή κάποιες αόριστες διατυπώσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν πολλά πράγματα, ούτε θα συνεισφέρει σε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιολάινεν. Ε, Ευχαριστώ, Νικολά, για την στράτευσή σου, τον ενθουσιασμό που είδαμε όχι μόνο στη διάρκεια της Λουξεμβουργικής Προεδρίας, αλλά βλέπω ότι σε διέπουν ακόμη. Ευχαριστώ λοιπόν είναι η δεύτερη μου προεδρία, η δεύτερη Λουξεμβουργική προεδρία, την οποία ζω προδεκαετία επίση. Σα είχα ξαναδεί. Ε, το Λουξεμβούργο λοιπόν είναι ένα ζωντανό και ενεργό εταίρο μέσα στην Ένωση, κάτι που δεν μπορώ να πω για όλε τι χώρε τη Ένωση. Περνούμε μέσα από κρίση, όντω. Δεν υπάρχει μονάχα έλλειψη αλληλεγγύη, υπάρχει και έλλειψη πειθαρχία και πίστη στο δίκαιο, στι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί προβλέπουν ακόμη ότι μπορεί και να καταρρεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν προσέξουμε. Πάντως η κατάσταση όντως διαμορφώνεται σοβαρή και αν συνεχίσουμε τα πράγματα έτσι όπως ε, ε, διεξήχθησαν κάποια πράγματα στη δική σας Προεδρία αρχίζουμε να απομακρυνόμαστε. Εγώ θεωρώ πάντως ότι κάποιοι θεσμικοί ε, κάποια, κάποιοι θεσμοί μάλλον λειτουργούν, αποδίδουν. Κομισιόν, Κοινοβούλιο λειτουργούν ω θεσμοί. Ο αδύναμο κρίκο είναι το Συμβούλιο. Πώ μπορεί κανεί να βελτιώσει τη λειτουργία του Συμβουλίου. Σε αντίθεση με τον αγαπητό Σέπφριν, δεν θα πω ότι απόφαση κατά πλειοψηφία σημαίνει δικτάτ. Γιατί αν το δεχτούμε αυτό, α ξεχάσουμε οποιαδήποτε πολιτική τη Ένωση. Υπάρχουν ψηφοφορίε και αποφάσει κατά πλειοψηφία. Το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει κατά πλειοψηφία. Συνήθω αναζητεί την ομοφωνία, κάτι το οποίο είναι και καλό είναι και κακό. Συνήθω δηλαδή και αργεί και καταλήγει σε ένα χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Μήπω θα πρέπει το Συμβούλιο να δείξει περισσότερο θάρρο και να λάβει περισσότερε αποφάσει κατά πλειοψηφία. Έχω και το άλλο διαρκέ ερώτημα του τρόπου επικοινωνία από πλευρά μα ω Ευρωπαϊκή Ένωση προ την κοινή γνώμη. Βρισκόμαστε στον, στον αιώνα των κοινωνικών μέσων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κατακυριεύουν τον κόσμο και εμείς ακόμα λειτουργούμε με ανακοινοθέντα τύπου. Κάτι που να κάνουμε εκεί, διότι δεν φτάνουμε στα όματα της κοινή γνώμης, ενώ οι αντίπαλοι του σχεδίου ολοκλήρωσης της Ευρώπης βασίζονται πολύ στα ε, κοινωνικά μέσα είχε υπάρξει και η πρωτοβουλία Debate Europe με την ε, κυρία Μάλμστρομ τότε πρωτοδεκαετία. Πού προχώρησε, πόσο προχώρησε αυτή. Σας ευχαριστώ τώρα για την υποστήριξή σας για την ε, μεταρρύθμιση του εκλογικού δικαίου. Συναντηθήκαμε με το Κορεπέρ και ο Βρετανός πρέσβης μας είπε ότι ούτε ένας Βρετανός Ευρωβουλευτής δεν υπερψήφισε. Και ο Δανός είπε «Α, και οι δικοί μου απέσχον». Όμως οι συνάδελφοί μας ψήφισαν υπέρ σε πολλά θέματα. Στο τέλος, στην τελική ψηφοφορία, είχαν κάποιες δυσκολίες ορισμένα από τα θέματα και γι' αυτό είτε καταψήφισαν είτε απέσχον. Υπάρχουν όμως άλλα θέματα που συγκεντρώνουν ευρύτατες πλειοψηφίες. Δεν αποτελεί αυτό βέβαια δικαιολογία για ορισμένες ε, χώρες μέλη που κινούνται αντίθετα με το ρεύμα. Οι εκπρόσωποι όμως, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των ε, χωρών αυτών ψήφισαν μαζί μας σε πολλά σημεία, όχι όμως στην τελική ψηφοφορία, αυτό το επισημαίνω, έχει σημασία. Ευχαριστώ. Ραμόν. Καλησπέρα, Υπουργέ. Να σας καθησυχάσω, δεν πρόκειται να σας μιλήσω για την Εξεταστική Επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερος προσωπικά εσάς για την δουλειά σας. Να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο ανοίξατε μια οδό που ελπίζουμε να την διατάξουν κι άλλοι. Μια και κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση εδώ και μια και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε έτσι, θα ήθελα να σας μιλήσω για ότι συμφωνώ με αυτή την Ευρώπη των αξιών. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Σμιτ, αλλά θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο είπε και ο Γιολάινεν. Σχετικά, σχεδόν όλα όσα έχουμε στα χέρια μας, τελικά ε, προσκρούει στην αντίρρηση του Συμβουλίου. Το βλέπουμε αυτό στο Κοινοβούλιο. Όταν στρέφουμε προς τα πίσω, ε, Είδα και άλλα σημεία και άλλες στιγμές χρονικές στην ε, ευρωπαϊκή οικοδόμηση, όχι τόσο μεγάλες όπως αυτή που ζούμε τώρα, γιατί σαφέστατα ζούμε ε, μια πολλαπλή κρίση οικονομική, το Brexit, το Brexit, τον τρομοκρατία, τους πρόσφυγες, σαφέστατα. Αλλά υπήρξαν και άλλες ε, περίοδοι στην περίπλοκη ιστορία της Ευρώπης, όπου υπήρχε ένα ρεύμα, μια τάση, όπου τα κράτη, όχι η Κομισιόν, μόνο, ούτε μόνο το κοινοβούλιο, τα κράτη πήγαν, πήγαιναν προς μια κατεύθυνση και είχαν την ικανότητα να προχωρήσουν προς τα εμπρός, να βρουν λύσεις. Η συνθήκη της Λισαβόνας, μεταξύ την αποτυχία που είχαμε με τα δημοψηφίσματα στην Γαλλία και στην Ολλανδία, ε, που δημιούργησαν τροχοπέδι στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Αλλά μην ξεχνάτε την, την το Μάστες κτλ σας μιλάω για αυτή την αίσθηση που έχω, έτσι, και το λέω με κάθε ζεστασιά, είναι ότι το Συμβούλιο κάνει ενδογαμικού τύπου προσπάθειες. Τα κράτη δεν έχουν αυτή τη διάθεση για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Παρότι ότι όλα αυτά που συμβαίνουν απαιτούν περισσότερη Ευρώπη. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Φέτος είχαμε μια κρίση δημοσιονομική άνευ προηγουμένου. Υπάρχει ε, ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα ε, λόγω της φοροαποφυγής με τα με τις φορολογικές συμφωνίες κτλ. Και σε τέτοιες κρίσεις οι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι πλώσαν πολύ για την κρίση. Μέσα σε αυτή την κοινωνική έτσι, ανησυχία έχουμε το Μοσκοβισί που μας, δημιουργείται, μας ότι δημιουργείται μια ειδική επιτροπή ε, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια καλύτερη, ένα καλύτερο συντονισμό ε, για τα δημοσιονομικά που προσκρούμε στο Συμβούλιο. Όπου λέει ότι δεν, μπορεί να, δεν υπάρχουν αρμοδιότητε ούτω ώστε άλλοι ε, οι Κομισιόν ε, προκειμένου να κάνουν αυτό τον συντονισμό. Ο, όμως Κοβισή ήθελε ε, να γίνει μια συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με ειδικού κανόνε για τα δημοσιονομικά. Και η, η Κομισιόν θα ήθελε μόνο ε, έτσι, ένα ρόλο υποπτίας. Αλλά τα κράτη τι είπαν, όχι, δεν έχετε αρμοδιότητα. Σήμερα το πρωί ο Υπουργό Εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια δήλωση εδώ που μου φαίνεται πολύ σοβαρή εμένα. Γιατί έχει δίκιο. Έλεγε ότι αν υπήρχαν περισσότερε, αν ανταλλάσσαμε περισσότερε πληροφορίε στην καταπολέμηση τη δημοκρατία, μπορεί να είχαμε αποφύγει τι επιθέσει τις επιθέσεις στο Παρίσι. Σοβαρότατο μου φαίνεται αυτό, έτσι, γιατί είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ε, εδώ και δύο χρόνια Ζούμε μια πραγματικότητα τρομοκρατία στην Ευρώπη. Ξεκίνησε το 2004 στη Μαδρίτη. Μετά είχαμε το Λονδίνο κτλ. κτλ. Οι αστυνομικέ ε, αρχέ των ε, κρατών μελών δεν θέλουν όμω να μοιραστούν τι πληροφορίε και αυτό είναι ντροπή. Είναι απαράδεκτο. Και πού κολλάει το πρόβλημα, πού προσκρούει στο Συμβούλιο Ποιο δεν θέλει μια ευρωπαϊκή αστυνομία που θα, αναλύει, που θα συντονίζει την πληροφορία. Ποιο δεν θέλει το Συμβούλιο. Αυτή είναι η ερώτησή μου και ζητώ συγγνώμη για αυτή την έντονη έκφρασή μου. Οι εκάστοτε εξαμηνιές προεδρίες ή η δικη σας ή ε, μια μόνιμη προεδρία, γιατί πριν από τρεις μέρες ο κύριος Τούσκ πήγε στην ε, Σοσιαλιστική Κοινοβουλευτική Ομάδα για να μιλήσει και με απογοήτευσε πλήρως. Σας ρωτάω λοιπόν, υπάρχει πολιτική ηγεσία εδώ πέρα. Το Συμβούλιο ξέρει που πάμε. Υπάρχει συντονισμό για αυτή την ε, προβληματική Ευρώπη που βρίσκεται σε κρίση. Δεν θέλω να σας επιπλήξω τώρα. Είναι ένας προβληματισμός που κάνω μεγαλόφωνα. Ε, bon, je, je, je comprends tout. Κατανοώ ότι ο πρώτος που κατηγορείται είναι το Συμβούλιο. Ανήκω στο Συμβούλιο. Ακόμα και αν δεν το εκπροσωπώ πλέον άμεσα. Το Συμβούλιο αντικατοπτρίζει τις αντιφάσεις μεταξύ κρατών μελών. Είναι ξεκάθαρο. Έχετε αντιφάσεις. Σας το λέω ειλικρινά. Υπάρχουν και εδώ αντιφάσεις. Υπάρχουν κάποιοι που εκφράζουν απόψεις που δεν τις συμμερίζονται όλοι. Και είναι και υπερβολικές ε, λοιπόν, ε, έχω μάθει να ακούω εδώ και μερικούς μήνες αυτές τις θέσεις. Αυτό που αναφέρατε για μια κοινή θεώρηση των πραγμάτων. Πέρα από τις διαφορές. Αυτό το κοινό όραμα ε, τελικά διαλύεται και αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Εγώ είπα ότι η αλληλεγγύη πρώτα απ' όλα είναι η διάθεση είναι μια θεμελιώδης προσέγγιση. Αυτή είναι μια πολύ βασική αρχή. Αν αρχίζουμε να σχετικοποιούμε τις θεμελιώδεις αρχές και πάμε προς μια προσέγγιση ο καθένας για τον εαυτό του, δεν πρέπει να εκπλησόμεθα που αποδυναμώνεται η Ευρώπη. Όλα τα κράτη-μέλη, όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί θα πληρώσουν το τίμημα, πολύ μεγάλο τίμημα, αν γίνει αυτό. Αυτή είναι η βραχυπρόθεσμη πολιτική και έχουμε και την πολιτική που χρειάζεται μακρόπνοη θεώρηση των πραγμάτων. Ίσως αυτό να λείπει σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Για την ψηφοφορία, την ψήφο με πλειοψηφία είναι μια αναγκαιότητα. Αν πρέπει να υιοθετούμε τα πάντα με ομοφωνία ακόμα και σε κάποιους τομείς, τομείς πρέπει να το κάνουμε, προβλέπεται ομοφωνία, αναφέρθηκε ένας τομέας, η φορολόγηση, δεν θα προχωρήσουμε. Δεν θα προχωρούμε το ρυθμό που απαιτείται, γιατί ο κόσμος προχωρά. υπάρχουν εξελίξεις, προχωρούν οι εταιρείε. Και η Ευρώπη πάει με το ρυθμό που υποχρεούται να πάει και άλλοι κινούνται με ταχύτητα του φωτός. Επιταχύνει η τεχνολογία τα πάντα σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ψηφοφορία με την ειδική πλειοψηφία, να εξασφαλιστεί αυτό, ακόμα και αν κάθε φορά προσπαθούμε να βρούμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Φτάνει η στιγμή όμως που πρέπει να ψηφίσει κανείς με ειδική πλειοψηφία όταν το προβλέπουν συνθήκες. Αν το προβλέπουν συνθήκες, γιατί να μην το εφαρμόσουμε. Δεν θα εφαρμόζουν πλέον τις συνθήκες. Δεν είναι τιμωρία να είναι κανείς στη μειοψηφία. Είναι μια δημοκρατική αρχή. Πρέπει κανείς να δέχεται καμιά φορά στη μειοψηφία. Και η βασική αλληλεγγύη που η του εχειρήματο Ευρωπαϊκού είναι αυτό. Να δέχεται κανείς ότι μπορεί κάποτε να μπει στη μειοψηφία και θα πρέπει να εφαρμόσει αυτά που αποφασίζει η πλειοψηφία. Αυτή είναι η κοινή κυριαρχία. Αλλιώ να θέτει κανεί την κυριαρχία του στην κοινή απόφαση. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Όσον αφορά τη συζήτηση για την Ευρώπη, Ε, ε, είμαι παλιός εγώ εδώ, τα ξέρω αυτά όσον αφορά τη συζήτηση για την Ευρώπη, επικοινωνία για την Ευρώπη, Communicating Europe. Ένας Ολλανδός συνάδελφος είχε την πρωτοβουλία για την Ευρώπη, την επικοινωνούσα. Θα πρέπει ο καθένας εκεί που βρίσκεται, εκεί που έχει τις ευθύνες, να κάνει τη δουλειά του για να συζητεί, να πείθει, να επικοινωνεί, να προωθεί την Ευρώπη. Τώρα, να επεξεργαστούμε μεγάλες ε, στρατηγικές και να δώσουμε χρήματα σε εταιρείε επικοινωνιών και να πουλάμε την Ευρώπη όπως πουλάμε άλλα προϊόντα, οποιοδήποτε προϊόν, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό θα δουλεύει και όλο λιγότερο πείθομαι. Όσο πουλάτε τόσο πιστεύει ο κόσμος, θα πρέπει να πείθετε. Να πείθετε και με την πρόοδο. Διότι γιατί υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης. Η κρίση εμπιστοσύνης υπάρχει διότι ίσως τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα στο απαιτούμενο ύψος. Το είπαν κάποιοι αυτό. Πρέπει να πείθουμε για να δείξουμε ότι χωρίς την Ευρώπη κολλάμε, πέφτουμε στον τοίχο. Σε πολλά θέματα. Και σε άλλα θέματα θα προχωράμε αλλά θα υποχωρούμε. Είναι θέμα επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αστυνομία, αυτά που είπατε, συμφωνώ. Δεν πρέπει εξ αντιδράσεως να λέμε ότι δεν θα επικοινωνούμε. Δεν είναι απαντήδες που υπάρχει επικοινωνία. Είναι θέμα νοοτροπίας. Στις νομικές δυνάμεις μπήκαν σχετικά αργά στις νομικές δυνάμεις στη λογική την ευρωπαϊκή. Το Μάστριχτ. Είχαμε την Τρέβη πριν λοιπά, Αλλά δεν ήταν τόσο επίσημο. Το Μάστριχτ για πρώτη φορά δημιούργησε τη δική δικαιοσύνη εσωτερικών κλπ είναι ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί, θα πρέπει να βελτιωθούν τα δίκτυα και να υπάρχουν πραγματικά τα αντανακλαστικά. Να πούμε, ιδού μια πληροφορία πρέπει να μοιραστεί σε όλους. Εδώ κοντά συλλάβαμε κάποιο στα σύνορα. Αν η γαλλική αστυνομία είχε τις πληροφορίες που είχαν οι βελγικές αστυνομικές αρχές, αυτό το άτομο θα είχε συλληφθεί και η γαλλική αστυνομία δεν είχε τι πληροφορίε. Νομίζω ότι αυτά τα δραματικά, τραγικά γεγονότα θα έπρεπε να είναι πραγματικό μάθημα. Να πούμε ότι δεν πρέπει πλέον να το δεχόμαστε αυτό, να μην ανεχόμεθα τέτοια κενά. Τώρα για τη φορολόγηση, εγώ είμαι λιγότερο απεσιόδοξο από εσά. Γνωρίζω αρκετά καλά το θέμα αυτό και γνωρίζω ότι έχουν επιτευχθεί κάποιες πρόοδοι. Αυτά που κάναμε τους τελευταίους μήνες τα δύο τελευταία χρόνια ας πούμε, δεν θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε εδώ και κάποια χρόνια. Ε, νομίζω ότι υπάρχει μια βούληση από αυτού η φορολόγηση να προχωρήσει. Βεβαίως υπάρχουν κάποια κολλήματα, πρέπει να το δεχτούμε, όσον αφορά το θέμα αυτό, το προοδικό τουλάχιστον, υπάρχει πρόοδος ε, και στα οικονομικά εντός της ενώσεως, διότι ίσως και σε διεθνή κλίμακα εξελίσσονται τα πράγματα. Έχουμε τη μία πλευρά την πτυχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και από την άλλη πλευρά έχουμε όλα αυτά που γίνονται σε άλλους χώρους, στον ΟΣΑ, Φερρυπίν, όπου και εκεί κινούνται προς μια συνεργασία για τα φορολογικά, καταπολέμηση κάθε είδους ε, φόρο διαφυγή και φοροαπάτη, κάτι που δικαιολογείται. Ίσως τα κράτη καταλαβαίνουν ότι αν θέλουν να επιβιώσουν οικονομικά δεν μπορούν να παίζουν το παιχνίδι της διαφυγής ο ένας ή μια χώρα κατά της άλλης. Και για τη συζήτηση για την έκθεση της Μεσάντες Μπερσόν και Τέλμαν Μπροκ. Η ιδέα τη συνεδριάση του, κοινωνικού, του Συμβουλίου Κοινωνικών Θεμάτων για την Ευρωζώνη, τι έγινε. Απάντηση. Ελπίζω να μην εξαφανίστηκε αυτή η ιδέα. σαν εκπρόσωπος κράτους μέλους μαζί με άλλους θα το προωθήσω. Είχε επικριθεί από κάποιους, είχε υποστηριχθεί από κάποιες χώρες. Είναι κάτι που πρέπει να το επεξεργαστούμε, Ίσως να βρούμε πιο εύκαμπτες λύσεις. Οργανώσαμε το Eurogroup επί της βάσης στην, στην ίδια μορφή που είχε και το οικονομικό Eurogroup κάποιο τμήμα το Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ θα πρέπει να ασχολείται με κοινωνικά θέματα που αφορούν άμεσα τις χώρες της Ευρωζώνης ή τους διάφορους μηχανισμούς του ευρώ, αλλά όλα τα κράτη-μέλη που επιθυμούν μπορούν να παρίστανται. Διότι γνωρίζω ότι έχουμε κάποια κάτι μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, που δεν θέλουν να διαχωριστούν από την κοινωνική πρόοδο, θέλουν να ανήκουν στην κοινωνική πρόοδο ακόμα και αν δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να βρούμε κάποιες λύσεις ενδεδειγμένες, είναι σημαντικό όμως η κοινωνική διάσταση να λαμβάνεται υπόψη. Κάναμε κάποια πρόοδο σχετικά με αυτό στην Προεδρία μας. και να λαμβάνεται υπόψη κοινωνική διάσταση στην οικονομική διακυβέρνηση. Και ευχαριστώ και το Κοινοβούλιο για τι εκθέσει του σχετικέ. Να συνεχίσω, Ρε Πρόεδρο. Εξαρτάται από το Συμβούλιο να ξεκινήσει τι εργασίε για την δημιουργία αυτού του φορολογικού συμφώνου και να ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είπατε ότι πρέπει να εξετάσουμε και τον κοινωνικό πυλώνα, όπω αποκαλείται. Δεν έχει ξεκινήσει προβληματισμό στο Συμβούλιο. Απάντηση. Αυτό είναι ένα τμήμα της συζητήσεως που στρέφεται γύρω από την έκθεση των πέντε πρόεδρων. Και θέλουμε να δούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να προοδεύσουμε όσον αφορά την εμβάθυνση τη ευρωζώνη. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται. Δεν θεωρείται σαν πρώτο βήμα το πρώτο βήμα που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δεύτερο βήμα που προτάθηκε δεν προβλέπει καμία αναθεώρηση των συνθήκων. Ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με αναθεωρήσεις των συνθήκων. Γνωρίζουμε όμως ότι πιθανότατα εάν θέλουμε εμβάθυνση και ενίσχυση της Ευρωζώνης θα πρέπει να προβούμε και σε κάποιες μεταρρυθμίσεις των συνθήκων. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι δεν είναι ιδιωτικό σχόλιο, ότι θα μας λείψετε. Δεν έχουμε τόσους υπουργούς στην Ευρώπη με τέτοια θεσμική μνήμη, αφοσίωση, κατανόηση, πάθος, όραμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν χαρά που εργαστήκαμε μαζί σας, συνεργαστήκαμε. Χαρά δική μου λέει ο κ. Υπουργός και αποχωρεί. <laughs> Now we can move... Τώρα, α ναι, θα περιμένω να αποχωρήσει ο κύριος Υπουργός.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 Θα μείνω και μαζί σας άλλωστε. Ας δώσουμε αμέσως το λόγο τότε. Ή να περιμένουμε λίγα λεπτά. Ό,τι θέλετε. Μπορούμε, μπορώ να είμαι πολύ σύντομη γιατί είμαστε όλοι και όλοι τρεις εδώ λέει η κυρία Μπρέσο. Ε, βέβαια, κοιτάξτε, είναι και, είναι και πέμπτη απόγευμα, είναι το πρόβλημα γνωστό. Α, είναι όμως κανονική ημερήσια ε, εργάσιμη ημέρα, λέει η πρόεδρος Χιούπνερ. Ωραία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε λίγοι, αλλά παθιασμένοι με το θέμα. Προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γιατί έχουμε ήδη αναφέρει τις αρχές που μας ε, καθοδήγησαν για την σύνταξη αυτού του εγγράφου. Όχι μόνο μία φορά, αλλά δύο-τρεις φορές και οι ακροάσεις μας, ας πούμε, στην Κομισιόν και αυτές μας βοήθησαν. Θα υπενθυμίσω τους λόγους, λοιπόν, που μας κάνουν να συντάσσουμε την, την έκθεση. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις σημαντικές, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από τα κράτη-μέλη. Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλονιστεί. Πρέπει να προσπαθήσουμε για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια των θεσμικών οργάνων και να δείξουν τα θεσμικά όργανα μεγαλύτερη ικανότητα να ολοκληρώσουν το έργο τους. Είμαστε πεπισμένοι ότι στο εσωτερικό της συνθήκης της Λισαβόνας υπάρχει ένα δυναμικό πολύ σημαντικό που δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα και πολλά από τα εργαλεία που υπάρχουν στην συνθήκη της Λισαβόνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουμε αυτές ακριβώς τις προκλήσεις. Η κοινωνική μέθοδος είναι ανώτερη από τη διακυβερνητική μέθοδο. Το αναφέραμε και πριν από λίγο. Και θα πρέπει να γίνεται πάντα σεβαστή και να χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο Χρησιμοποιώντα και όλα τα εργαλεία που υπάρχουν στο εσωτερικό συνθήκη συνθήκης Λισαβόνα και μας επιτρέπουν να περάσουμε από την ε, ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία για μία σειρά από θέματα. Όπως είπαμε πολλές φορές, η έκθεση εξετάζει καταρχάς τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στο εσωτερικό της λειτουργίας διαφόρων θεσμικών οργάνων Μιλάμε για το διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και γι' αυτό έχουμε μιλήσει εδώ στην συνεδρίασή μας. Να αυξήσουμε τη συνεργασία, αλλά σεβόμενοι ο ένας τις θεσμικές αρμοδιότητες του άλλου. Υπάρχει και ένα τμήμα αφιερωμένο στο Συμβούλιο. Μόλις αναφερθήκαμε στο θέμα του Συμβουλίου με τον Λουξεμβουργέζο Υπουργό. Το Συμβούλιο είναι ένας από τους αδύναμους κρίκους της λειτουργίας των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Έχει μια τάση να παίζει και ένα νομοθετικό ρόλο που δεν αναφέρεται όμως και δεν προβλέπεται στις συνθήκες και θεωρούμε ότι αν θέλει να έχει και νομοθετικό ρόλο, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη ρήτα της πασαρέλας για να περάσει από την, πλειοψηφ... από την ομοφωνία σε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία. Αντίστοιχος προβληματισμός, αλλά με πιο λεπτομέρειες, γίνεται ε, για το Συμβούλιο, πέρα από το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που στο εσωτερικό των συνθήκων μπορεί να μετασχηματιστεί σε μια πραγματική νομοθετική σε ένα πραγματικό νομοθετικό σώμα, αυξάνοντα τη διαφάνειά του, χρησιμοποιώντα. πολλά από τα τεχνικά συμβούλια ε, και φτιάχνοντας μορφώματα συμβουλίου ε, πιο νομοθετικού χαρακτήρα. Αυτό το ανέφερε και η συνταγματική συνθήκη αλλά τελικά αυτή η ρήτρα δεν πέρασε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν υπάρχει όμως, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιώντα του κανόνε που υπάρχουν στην συνθήκη της Λισαβόνα, αφού υπάρχει η σχετική θέληση. Δεν θα να Μιλάμε όμως και για το πρόβλημα της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου στην εκλογή των προέδρων της, του Προέδρου της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια σταθεροποίηση της διαδικασίας που εφαρμόστηκε την τελευταία φορά, αλλά που δεν είναι πάγια. Θα θέλαμε να δημιουργηθεί επίσης μια φορολογική διοίκηση και ένα ευρωπαϊκό ε, Υπουργείο Οικονομικών και να υπάρχει μια εκπροσώπηση Ευρωζώνης στα διεθνή φόρουμ. Επίσης ένα τμήμα αναφέρεται στην σωστή εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας. Η αρχή αυτή δεν είναι βάρος, είναι ο σεβασμός μιας Ευρώπης η οποία έχει οικοδομηθεί δίδοντας αρμοδιότητα στην Ένωση, αλλά κασταλίζοντας και το σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των υποεθνικών επιπέδων που εκπροσωπείται από την Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και την Ευρωπαϊκή και Οικονομική Επιτροπή. Υπάρχει μια οριζόντια επικουρικότητα, δηλαδή η ελεύθερη οργάνωση της κοινωνίας. Υπάρχει, υπάρχουν και μια σειρά από σκέψεις για την εμβάθυνση της ΟΝΕ. και μια νομική πράξη θα έλεγα για την οικονομική πολιτική της ε, ναι. μια απλούστευση και δημοκρατικοποίηση της ε, διαδικασίας που αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δεν θα το μακρηγορήσω γιατί είναι σαφές ότι αυτό που ήθελα να υπενθυμίσω σε μένα και στους συναδέλφους είναι ένας κατάλογος πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να φτιάξουμε αυτό το Ever Closer Union ε, που παρότι δεν του αρέσει του Κάμερον, σε εμάς μας αρέσει. Σε μας αρέσει και σε πολλούς άλλους στην Ευρώπη. Δεν αρέσει σε όλους τους Ευρωπαίους, αλλά σε πολλούς Ευρωπαίους αρέσει. Προτείνουμε επίση να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τον προϋπολογισμό της Ένωσης, να βελτιώσουμε τον τρόπο ψηφοφορίας και των αποφάσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να αυξήσουμε την δυνατότητα επενδύσεων τη ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντα όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές σε όλους, ότι χωρίς αύξηση του, δυναμικού, του επενδυτικού τη Ευρωπαϊκής Ένωση, πολλά από τα πράγματα που περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν πρόκειται να γίνουν. Το θέμα της εσωτερική αγοράς, της υλοποίησης μιας πραγματικής φορολογικής ένωσης, ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο και, έτσι, και, μια, και αρχιτεκτονική για την ΟΝΕ. Και μπορούμε ακόμα και στο εσωτερικό της Λισαβόνας να τα καταφέρουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, να φτιάξουμε μια κοινωνική διάσταση. Εδώ έχουμε δύο προτάσεις. Υπάρχουν και πολλές άλλες, αλλά να υπενθυμίσω μόνο αυτές. Ε, ζητάμε από την Κομισιόν να δημιουργήσει ένα, μια δέσμη κοινωνικών κριτηρίων για να αξιολογούμε τις επιδόσεις στα κοινωνικά θέματα των κρατών μελών και θέλουμε να πάμε προς μια πραγματική κοινωνική συμφωνία που θα διασφαλίσει και θα επανεκκινήσει την κοινωνική οικονομία της αγοράς που από πάντα ήταν χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μακρύ τμήμα για προφανείς λόγους αφιερώνεται σε πολύ επίκαιρα θέματα που αντιμετωπίζουμε στην εξωτερική δράση, στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και δημοκρατικότητα της, των κοινών μας δράσεων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Ζητάμε από το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει τη ρητά της Πασαρέλας για να περάσει από την ομοφωνία εκεί όπου γίνεται σε λήψη των αποφάσεων και ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία. Να χρησιμοποιήσουμε την μόνιμη διαρθωμένη συνεργασία, αυτό το εργαλείο, για να πάμε προς την κοινή άμυνα στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποια πράγματα που κινούνται σε επίπεδο κομισιών. Θέλουμε να υπάρχει μια κοινή ακτοφυλακή. Μας άρεσε αυτή η πρόταση που έκανε η Κομισιόν για να ενισχύσουμε τη δράση των κρατών μελών. Και φυσικά σε ό,τι αφορά την πολιτική δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων, τζάι, το θέμα της διαχείρισης του περίπλοκου θέματος των προσφύγων, εδώ μπορεί να εξυπηρετηθεί από μια κοινή εκταφλάκη που είπα πριν και θα πρέπει ούτως ή άλλως να υπάρχει συντονισμό των ε, ευρωπαϊκών υπηρεσιών ε, πληροφοριών που πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται οι με τις δε. Λίγα, δεν ανέφερα όλα όσα λέει η έκθεση, λίγα ανέφερα. Παρ' όλα αυτά είπα αρκετά. Αλλά Πιστεύω ότι καταφέραμε να δείξουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολλά πράγματα χρησιμοποιώντας την ισχύουσα συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίε για να μην προχωρήσουμε γιατί δήθεν θα πρέπει να αλλάξουμε τη συνθήκη. Όχι. Αυτά είναι κάποια από τα πράγματα ε, που είναι σημαντικά και μπορούν να γίνουν στο εσωτερικό της συνθήκης της Λισαβόνας. Τα ζητάνε και οι εφημερίδες, οι δημοσιογράφοι κτλ νομίζω ότι είναι ένα ενθύμιο που μπορούμε να δώσουμε εμείς η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στα άλλα θεσμικά όργανα, στους ε, πολίτες που καθημερινά λένε «Α, η Ευρώπη δεν κάνει αυτό, δεν κάνει αυτό, πρέπει να το κάνει» ε, ή «Δεν πρέπει να κάνει το, το άλλο ας πούμε, που κάνει». Ε, να την μπορούμε να τους προσφέρουμε λοιπόν. Ε, you, you want to gegen diese volle Gewalt der Δεν έχω μετά από αυτόν τον οριμαχδό λέξεων να προσθέσω πολλά άλλα πράγματα διότι η Μεσέντες Πρέσο τα είπε όλα. Νομίζω πάντως συνεχίζει ο ο Μπροκ, ότι μπορώ να προσθέσω και αυτό είναι η προσωπική μου αντίληψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται βαθιά στην πιο σοβαρή κρίση της ιστορίας της. Είμαι ήδη 35 και πλέον χρόνια ευρωβουλευτής και για πρώτη φορά με διακατέχει το συνέστημα ότι το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μπορεί και να αποτύχει. Για πρώτη φορά και ότι καλούμαστε να διαπιστώσουμε ότι καμιά φορά δικαίως, καμιά φορά αδίκως και είτε αντικειμενικά είτε υποκειμενικά τα φορτώνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οφείλουμε νομίζω να φροντίσουμε να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Διαπιστώνω εξάλλου ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη σε πολλούς τομείς όσο μας εμποδίζει η αρχή της ομοφωνίας του δικαίου των συνθήκων και ότι σε αυτό το σημείο δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση της συνθήκης. Ως Ευρωπαίος Φεντεραλιστής θα ήθελα να δω νέο σύνταγμα που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει γιατί θα κολλήσει στη διαδικασία κυρώσεων από τις Εθνικές Βουλές. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση όπου ίσως έχουμε μια δυνατότητα να διατηρήσουμε τα κεκτημένα μέχρι ότου κατορθώσουμε να δείξουμε επιτεύγματα στους τομείς που απασχολούν τον κόσμο και που αυτά τα επιτεύγματα να τα εκτιμήσει δεόντως το σώμα των ψηφοφόρων. Όταν βλέπω ωστόσο ότι οι χώρες μέλη δεν ασχολούνται πλέον πώς μπορώ να συμβάλλω, δεν, θεωρεί, δεν εξετάζει κάθε φορά πώς μπορεί να συμβάλλει σε μια κοινή λύση, αλλά πώς μπορεί να αποσυνδεθεί από το σύνολο των υπόλοιπων. Διερωτώνται οι θύνοντες πώς μπορώ να φορτώσω τα δικά μου σφάλματα στην Ευρώπη. Και ότι αυτό το βλέπει κανείς παντού. Σε όλες σχεδόν τις χώρες μιλή. Ακόμα και σε χώρες όπου εγώ δεν θα το περίμενα λόγω της ιστορίας τους. Αυτά μας οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Από την άλλη μεριά οφείλω να πω ότι οι εναλλακτικέ που προτείνουν είτε από δεξιά είτε από αριστερά είναι ανύπαρκτες. Ουδής προχωρεί στην κατάθεση μιας πραγματικής εναλλακτικής προτάσεως. Όλοι μέμφονται Ουδής λέει τι θα πρέπει να γίνει. Αν όμως κάποιος έρχεται και θέλει να καταστρέψει, χωρίς να δώσει μετά μια συνέχεια, να κάνει το επόμενο βήμα, αυτό δεν έχει παρά μόνο καταστρεπτικό χαρακτήρα. Καθαρό ε, ρητό του Ρίτσαρντ Μπέρκ από τον οποίο ξεκίνησε ο συντηρητισμό. Αυτή πάντω είναι η δική μου νοοτροπία. Αυτά που βλέπουμε και αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε με τις Πρέσο και εγώ στο έγγραφό μας είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό να εξασφαλίσουμε περιθώριο δράσεων για το ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να τροποποιήσουμε το πρωτογενές δίκαιο των συνθήκων. Περιθώριο δράσεων για την επίλυση προβλημάτων. Αυτό σημαίνει περισσότερη χρήση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία. Πρέπει να δείξουμε ότι η μη προσφυγή στο μέσον αυτό οδηγεί σε μπλοκάρισμα και όχι σε λύσεις. Αυξάνονται οι δυσχέρειες με την ομοφωνία. Διότι όλοι ζητούν περισσότερα με αποτέλεσμα να γίνονται πιο δύσκολες οι αποφάσεις και πιο δαπανηρές. μόνο με ενισχυμένη η πλειοψηφία, η οποία προσφέρει επαρκή ασφάλεια και για μεγάλους και μικρούς μπορεί να είναι ο δρόμος προς τα εμπρός. Το δεύτερο είναι πρέπει να μιλήσουμε για διαφάνεια. Είπε ήδη η Mercedes Πρέσο και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εξήγησε τα, των δύο νομοθετικών σωμάτων η Mercedes Πρέσο. Χρειαζόμαστε διαφάνεια και υπευθυνότητα στο Συμβούλιο Υπουργών ώστε να μην μπορούμε μετά να παριστάνουν οι κυβερνήσεις όταν επιστρέφουν στι πρωτεύουσέ του, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα υπόθηκαν ή αποφασίστηκαν στι Βρυξέλλε. Και αυτό πρέπει να καταστεί σαφέ μέσα από διάφανη κοινή συζήτηση. Και για μικρά πράγματα όπω αυτά που συζητούμε εδώ, στο Ευρωκοινοβούλιο. Η συνήθειά μα να προχωρούμε στη λήψη αποφάσεων. Με αδιαφάνεια είναι αυτή που οδηγεί σε απόσταση από τους πολίτες. Όταν είναι κανείς συγητής και προχωρεί σε μια συμφωνία που λύγει στην πρώτη ανάγνωση και δεν γίνεται επομένως ανοιχτή συζήτηση. Ανοιχτή συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αλλά ούτε και ανοιχτή συζήτηση μέσα στο ίδιο το Κοινοβουλίο. Πώς θα κατανοήσει εν τέλει ο πολίτης για ποιο λόγο είναι αναγκαία η νομοθεσία αυτή. Έρχονται οι εισηγητές και δείχνουν την ισχύ τους όπως θεωρούν ενώ μέσα στον κοινοβουλευτισμό προβλέπονται και δύο και τρεις αναγνώσεις ώστε ενδιάμεσα στις αναγνώσεις να μπορούν να διεξάγονται οι συζητήσεις με συμμετοχή όλων των διαφέρων μερών σε διαφάνεια στα όματα της κοινή γνώμης. Πράγμα το οποίο νομιμοποιεί τις τελικές αποφάσεις. Αλλιώς πέφτουν από τον ουρανό οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κεφάλια των ανθρώπων και βεβαίως αυτοί δυσαρεστούνται διότι δεν έχουν ιδέα Και γι' αυτό όργανα όπως το Συμβούλιο λειτουργούν σε αδιαφάνεια. Και οι συζητήσεις δεν διεξάγονται ανοιχτά ή πάντως όχι παρκώς με ανοιχτό κοινοβουλευτικό τρόπο. Γι' αυτό νομίζω μπορούμε να θεσπίσουμε ένα πρότυπο το οποίο πρέπει να καταστεί σαφές σε μια συζήτηση σε πολλούς τομείς από την εξωτερική πολιτική μέχρι την νομισματική και οικονομική πολιτική, τη δημοκρατική συμμετοχή, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και όλα αυτά στη βάση των γενικών σκέψεων που εξήγησα μόλι. Τα περιλαμβάνουμε όλα αυτά με πολλέ λεπτομέρειε. Δεν περιλαμβάνει πάρα, πολύ, πάρα πολλά νέα στοιχεία η έκθεση αυτή. Είναι η μετάφραση του working document και η μεταφορά των συζητήσεων που κάναμε το Δεκέμβρη μαζί με οι δήμονε και με εθνικά κοινοβούλια. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επαναλάβω όλες τις λεπτομέρειες. Πρέπει να δείξουμε και δυνατότητα ανάληψης δράσης ως Ευρωπαϊκή Ένωση και στο προσφυγικό και στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από τη συζήτηση αυτή. Μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Παρισιού επικαλέστηκε η Γαλλία το άρθρο 42 παράγραφος 7. Όλοι στην Κομισιόν και το Συμβούλιο έτρεξαν να δουν τι σημαίνει αυτό. Και διεπίστωσαν ότι πρόκειται για μια δράση διακρατική, όχι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπίστωσαν επίσης ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει κανένα συσχετισμός. Είναι σαν τον ενέργειο έχω αλλά ποιος κάνει το συντονισμό. Ενώ αυτό είναι το νόημα. Να μπορούν να υπάρχουν αυτόματοι μηχανισμοί οι οποίοι να διευκολύνουν τη συνεργασία των χωρών μελών. Μικρό παράδειγμα αυτό. Ακούμε διαρκώς μεγαλώσαμε διακηρύξεις και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και είναι πολύ δύσκολο μετά να βρει κανείς πού απολύγουν τα πράγματα αυτά στην πράξη. Αν δω τις αποφάσεις από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα για το θέμα των προσφύγων και των μεταναστών. Και ποια από αυτά έχουν εφαρμοστεί, ποια από αυτά έχουν εφαρμοστεί στην πράξη. Έχω δυσκολία να τα εξηγήσω αυτά. Διότι οι μηχανισμοί δεν αποδίδουν. Οι αποφάσεις είναι αδιαφανείς και δεν είναι και αποτελεσματικές διότι δεν εφαρμόζονται εν τέλει. Ας μην εκπλησώμεθα λοιπόν που οι πολίτες βγαίνουν και λένε δεν γίνεται έτσι δεν τα καταφέρνετε. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα σωστό. Αλλά αυτή είναι τελικά η εντύπωση. Στην πολιτική πραγματικότητα είναι μονάχα αυτή που διαμορφώνεται στα μάτια των πολιτών. Αν δεν κλείσουμε το κενό αυτό, αν δεν καλύψουμε το κενό αυτό, προχωρούμε σε μια πρώτη ως απώλεια αξιοπιστίας. Ευχαρίστω να συζητήσετε επιμέρους μαζί σας, αλλά δεν θέλω να σας λούσω περισσότερο ακόμα με όλη αυτή τη δυσαρέσκειά μου. Θεωρώ πάντως ότι τούτος εδώ ο χρόνος, ο καινούριος χρόνος, θα είναι μοιραίος για την Ευρώπη και λόγω επαπειλούμενου Brexit και λόγω αύξησης της εκλογικής δυνάμεως, ριζοσπαστικών δυνάμεων από δεξιά και από αριστερά Το να φανταστούν ορισμένοι ότι χορεύοντας με τους λύκους μπορούν να τους κρατήσουν μακριά, εκεί κάνουν μεγάλο λάθος. Μπορεί λοιπόν να αποβεί μοιραίο το έτος αυτό. Να δούμε λοιπόν αν σε τέτοια θέματα, όπου δεν είναι δυνατόν να γίνει η τροποποίηση της συνθήκης, παρόλα αυτά, στη βάση της συνθήκης αυτής, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε μεγαλύτερη διαφάνεια για να, μπορούσουμε, να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις που να εξυπηρετούν εν τέλει τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ξεκινήσει η συζήτηση. Ερωτήσεις μήπως. Προθεσμία για αποβολή τροπολογιών. Πότε είναι? 12 Φεβρουαρίου νομίζω. Ναι. Υπάρχει χρόνος για τις τροπολογίες. Υπάρχει και χρόνος σήμερα η συζήτηση. Πασκάρτηρο 12 το μήνος, 12 Φεβρουαρίου για τις τροπολογίες. Προθεσμία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύσκολο να πάρει κανείς τον λόγο μετά τη λαμπρή και πλήρη παρουσίαση που έλαβε χώρα το κάνω από σεβασμό προς τον Σβέν Γκίγκοντ που απουσιάζει σήμερα και μου έδωσε τις παρατηρήσεις του να σας διαβιβάσω. Ε, je crois ε, Ο Σβέν Giegold συμμερίζεται τα βασικά στοιχεία που έχουν γραφτεί και αναφέρθηκαν στην έκθεση, δεν την άκουσε, τη διάβασε. Αν άκουγε κιόλα, θα συμμεριζόταν τα σχόλια τα περισσότερα. Πρώτο σημείο στο οποίο ζητάει σας ζητά να επιμείνετε είναι η εργασία όσον αφορά τη ρήτρα Πασαρέλα και το άθρο 48 της συνθήκης επιτρέπει να περάσουν την ψηφοφορία σε, με ομοφωνία, σε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο. Προτείνει και επιμένει από αυτού ότι θα μπορούσαμε ίσως να καθορίσουμε ήδη κάποιους τομείς, ιδίως πόρους παραδείγματος χάρη, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, περιβαλλοντικές πολιτικές των κρατών μελών, που έχουν αντίκτυπο για την ενεργειακή πολιτική και επιλογή, γιατί ξέρετε θα επανέλθουμε στο θέμα της ομοφωνίας σε αυτά. Πάνω σε αυτά θα επιθυμούσε μια κάποια ευάθυνση όσον αφορά την έκθεση. Για το Eurogroup το θέμα της διαφάνειας του οργάνου αυτού του ανεπισήμου επιβάλλεται και τίθεται επιτακτικά και βάσει των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Αυξάνονται τα προνόμια και δεν υπάρχει έλεγχος. Τίθεται το ερωτηματικό λοιπόν και το ζήτημα. Και η έκθεσή σας έχει στόχο προφανώς να το καλύψει και αυτό. Όσον αφορά τους μεθοριακούς ελέγχους, Για το ΣΒΕΝ δεν τίθεται θέμα. Χρειάζεται η πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή διαχείριση από αυτού. Δεν θα σε εκπλήσει η θέση του ΣΒΕΝ. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε να επιμείνουμε στην εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των ετούντων άσυλο. Υποφέρουν, ε, βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Η έκθεσή σας αν μπορούσε να επιμείνει από αυτού και να καλύπτει την ανθρωπιστική πλευρά των ετούντων άσυλων, να λαμβάνετε υπόψη αυτή τη πτυχή πιο επίσημα, να τονίσετε περισσότερο. Θα ήταν έξοχο αυτό. Τελευταίο, που αναφέρθηκε τον κύριο Μπροκ, σαφέστατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την τρομοκρατία, την ασφάλειά της, έχει μείνει πίσω, ε, κυρίως πίσω όσον αφορά την ανταλλαγή ε, των πληροφοριών. Είδαμε ότι θα πρέπει να ε, γίνεται πιο εύκολη ανταλλαγή στοιχείων, κάτι που ζητούσε και η Γαλλία. Κυρίως όταν έχει επιπτώσει για την Ευρώπη. Όπως αυτή η παρέμβαση, η επέμβαση ε, του Γάλλου Υπουργού Εσωτερικών όταν αναφέρθηκε σε αυτό είπε ότι φταίει η Ευρώπη. Ενώ η Γαλλία και άλλες χώρες μπλοκάρουν συστηματικά, επανειλημμένα τις ανταλλαγές πληροφοριών. Θα ήταν καλό λοιπόν η έκθεσή σας να διευκρινίζει ότι το πρόβλημα το ευρωπαϊκό που τίθεται και κατά της εγκληματικότητας, οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας είναι πάνω απ' όλα ότι χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων χωρών και των διαφόρων μυστικών υπηρεσιών. Έλεγα το ίδιο και για θέματα δικαιοσύνη. Δεν στην έκθεσή σα. Βέβαια, γιατί είσαστε στο πλαίσιο των εθικών. Η ανυπαρξία στην Ευρώπη ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Ευρωπαίου Εισαγγελέα είναι προφανώ ένα μεγάλο, τεράστιο κενό όσον αφορά τη δυνατότητα να επεσπιστούμε ε, την Ευρώπη και ε, τις μυστικές, τη ε, συνεργασία μυστικών υπηρεσιών. Αυτά που μου ζήτησε ο Σβέν Γκίγκολτ να σας μεταβιβάσω και αυτό έκανα. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Ρίτσαρτ Κόρμπερτ, θες να πεις κάτι, θες να μιλήσεις. Ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της προθεσμίας για τις τροπολογίες. Πολιτικό ζήτημα ήταν περισσότερο, όχι πρακτικό η προθεσμία για τις τροπολογίες θα έπρεπε να περιμένει μέχρι ότου περάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Δεν ξέρουμε τι αποφάσει θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ίσως να λάβει κάποιες αποφάσεις συμπεράσματα που να επηρεάσουν αυτά που θέλουμε να πούμε εμείς στην έκθεσή μας και τι μπορούμε να κάνουμε εντό των πλαισίων των ισχυουσών συνθήκων. Πρόεδρος, θα προσπαθήσουμε. Θυμόσαστε πότε διεξάγεται το Συμβούλιο. 17-18. Χρειαζόμαστε τότε και μια εβδομάδα, να προτείνουμε μια εβδομάδα μετά και να δούμε και τι γίνεται με ψηφοφορία πότε θέλετε αυτό. Μπορούμε να το επενεξετάσουμε στο τέλος. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση της ουσίας. Γκέρολτ Φάνερμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους για τα όσα είπαν. Ευχαριστώ την κυρία Μπρεσό και τον κύριο Μπροκ για τις προτάσεις τους. Δεν θα σας εκπλήσει το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να διαφωνήσουμε περισσότερο. Αυτή είναι η θέση που θα υπερασπιστώ χωρίς να χρονοτριβήσω. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπρεσό που ήταν τόσο ανοιχτή και θερμή είπε ότι όλο και πιο στενή ένωση είναι κάτι που θεωρείται αυτονόητο και ξέρει ότι αυτό δεν αληθεύει για μένα. Ευχαριστώ τον κύριο Μπροκ, παρόλο που τον ευχαριστώ λιγότερο γιατί άρχισε να λέει ότι η άκρα δεξιά, οι ακροδεξιοί δεν έχουν εναλλακτική. Καταρχάς αυτό δεν αληθεύει. Επανειλημμένα υπογραμμίσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την βλέπετε εσείς είναι κάτι που δεν θα λειτουργήσει κατά την άποψή μας. Και η εναλλακτική είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία, όπου τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο και εξακολουθούν να έχουν ένα βαθμό αυτονομίας. Αυτό το έγγραφο εδώ μπροστά μας είναι ε, διαπνέεται από την ιδέα των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης ε, περιέχει φεντερλιστικά ιδεώδη ο κύριος Μπρόκ λέει ότι έχω την εντύπωση ότι όλα δεν είναι πλέον αυτονόητα. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι είπανε που είναι ο παλιός καλός καιρός όπου όλα ήταν πιο εύκολα και πιο αυτονόητα και όλοι κινούμεθα προς στην ίδια κατεύθυνση, την κατεύθυνσή σας δηλαδή. Δεν κινούνται όλοι προς την κατεύθυνση γιατί, διότι ε, δεν είναι οι ακροδεξιοί οι οποίοι συνομωτούν. Όχι, εσείς προχωρήσατε πολύ μακριά με την ολοκλήρωσή σας. Ξεπεράσατε πιο πέρα από αυτό που θέλαν οι Ευρωπαίοι πολίτες και κατά των ενδείξεων για το αντίθετο εξακολουθείτε να ακολουθείτε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έγιναν δημοψηφίσματα που ο λαό είπε όχι. Πηγαίνετε πιο αργά, με πιο αργό ρυθμό. Είχαμε εκλογέ και αμέσω μετά τι εκλογέ θυμάμαι την όλη ατμόσφαιρα που επικρατούσε. Σε πολλά κράτη-μέλη. Ο λαό απέρριψε την προσέγγιση, την οποία ακολουθεί και έκθεση. Αμέσω μετά τι εκλογέ φαίνεται να το είχατε καταλάβει αυτό. Όμως, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε τη θητεία μας, ακολουθήσατε ξανά άλλη κατεύθυνση. Έχουμε την έκθεση Verhofstadt, που προχωρεί περαιτέρω, ζητά μεταρρύθμιση των συνθήκων, αλλά ακόμα και αυτή η έκθεση πηγαίνει κατά, στέφεται κατά των αρχικών προθέσεων. Όλοι αμέσως μετά τις ευρωεκλογέ θεώρησαν ότι είχαν προχωρήσει πιο πέρα από ό,τι έπρεπε και κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας θα έπρεπε να αλλάξουμε κατεύθυνση. Όμως διαλύθηκε αυτή η ατμόσφαιρα. Και τώρα κάνετε σαν να μην τρέχει τίποτα και ότι όλα είναι ως συνήθως. Και ακολουθείτε μια θρησκευτική προσέγγιση προς αυτή την πορεία. Είστε ζηλωτής. Εγώ θα υποβάλω ε, τροπολογίες σαν θέμα αρχής ξέρω ότι δεν έχουν καμία σημασία συνήθως οι τροπολογίες μου και δεν επηρεάζουν την κατάσταση, αλλά ακολουθείτε σχεδόν θρησκευτική προσέγγιση. Ακολουθείτε κάποια ρητά, κάποιες υποθέσεις, κάποια δόγματα που δεν βασίζονται σε ε, πραγματικά στοιχεία, ούτε στα όσα δείχνει η κοινή γνώμη. Στην τελική σκέψη α λέτε ότι η κρίση των προσφύγων σε συνδυασμό με την τελική σκέψη β δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά από κάθε κράτο μέλος. Αυτό ίσως να είναι μια δήλωση στην οποία πιστεύετε με θρησκευτικό ζήλο, όμως δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει και είναι κρίμα το λέω αυτό σε μια αίθουσα γεμάτη από φεντεραλιστές, αλλά αυτή ακριβώς η συζήτηση γίνεται στα κράτη-μέλη. Μπορούμε να τα αφήσουμε όλα αυτά τα θέματα να τα λύσει η Ευρώπη ή όχι. Εσείς υποθέτετε ότι ναι έτσι είναι και είναι αυτονόητο. Η κοινοτική μέθοδος υπερτερεί, λέτε, στην τελική σκέψη ε, ε. Αλλιώς αυτό που θα έχουμε είναι κατακαιρματισμός, λέτε. Ε, ξανά, κινείστε βάσει της υποθέσεως ότι κινούμεθα προς τις Ηνωμένε Πολιτείες της Ευρώπης. Και φαίνεται να θεωρείτε ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι εξίσου καλή. Όμως, ξανά, η κοινή γνώμη έχει αντίθετη άποψη οι συζητήσει είναι ακόμα ζωντανέ που γίνονται σε κάτι μελη και δεν καταλαβαίνω πώ μπορείτε να κάνετε άλματα προ συμπεράσματα και να κάνετε κάποιε υποθέσει όταν γίνονται αυτέ οι συζητήσει. Το ίδιο ισχύει για την ε, ομοφωνία ή για τον κατακαιρματισμό. Ε, ή είπατε ομοφωνία ή κατακαιρματισμό, ομοφωνία ή τίποτα. Ε, γιατί να μην υπάρχει πιο διαμορφωμένη συμμετοχή όπως είχαμε και για το ευρώ αν κάποια κράτη-μέλη ε, συμφωνούν με κάποιες διατάξεις, με κάποιους κανόνες και άλλες χώρες δεν συμφωνούν, δεν είναι και το τέλος του κόσμου ε, και δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τα πάντα με την ειδική πλειοψηφία. Διαφορετικά η μόνη άλλη επιλογή είναι η ομοφωνία. Πάλι, σαν θρησκευτικό δόγμα το παρουσιάζεται, αλλά δεν ισχύει απαραίτητα. Στο ζήτα λατινικό λέτε ότι εκτιμώντας ότι οι προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μας δείχνουν ότι πρέπει να δημιουργήσουμε σταδιακά μια κοινή αμυντική πολιτική. Ξανά και εδώ. Γιατί. Μετά το διπλό α, η προσφυγική κρίση εκφράζει την ανάγκη για κοινή πολιτική για το άσυλο και την μετανάστευση. Αλήθεια, έχετε αποδείξεις περί αυτού. ξανά φαίνεται να θεωρείται ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν λέω ότι ε, ε, υπολείπεται από την, αυτό που λέτε από την αλήθεια. Ένα τμήμα όμως της δημοκρατίας είναι να ακούτε και τη μειοψηφία και να λαμβάνετε υπόψη και τις εξελίξεις και ποια είναι η άποψη του εκλογικού σώματος που σας ψήφισε. Δεν είναι ότι επειδή είμαστε μειοψηφία και δεν έχουμε την πλειοψηφία εμείς και επειδή εκείνοι που είναι επικριτικοί στο κοινοβούλιο δεν έχουν την πλειοψηφία και όλο και περισσότεροι είμαστε που επικρίνουμε ότι η πλειοψηφία πρέπει να μας αγνοεί. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό, να αγνοεί η πλειοψηφία τη μειοψηφία. Στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή ΑΦΚΟ, έχω ένα καθήκον. Καθήκον μου είναι να έχω μία φωνή διαφορετική, να εκφράζω διαφωνία. Φορολόγηση, φορολογική ένωση, κοινή στρατιωτική πολιτική, κοινή οικονομική πολιτική. Χρειάζεται κανείς κοινή οικονομική πολιτική, γιατί αυτό είναι άλλο λάθο που κάνατε. Το άλλο λάθος ποιο είναι, το ευρώ. Η κοινωνικο-οικονομική πολιτική μετά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία ούτε από αυτό. Για την ώρα αυτά έχω να πω και τα λέω αυτά εν είδη στις μελλοντικέ συζητήσεις που θα λάβουν χώρα αφού έχουμε τις τροπολογίες. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω περισσότερο μαζί σας. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να σας περιορίσω. Είμαι εδώ για να σας δώσω και το λόγο και εσάς, αλλά και να επιτρέψω στην πλειοψηφία που δεν σας αρέσει τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι συνέβη με τη μετάφραση. Εγώ δεν στείλετε σε εσάς όχι, όχι, όχι. Για το πώ λειτουργεί η Επιτροπή μιλάω. Όλοι έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν. Και εγώ, λέει ο, ο Ευρωβουλευτής, έχω το δικαίωμα επίσης ε, να μιλήσω και θα, θα κάνω χρήση αυτού του δικαιώματος. Πολύ σύντομα. Ο επόμενο ομιλητής. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κύριο Μπρόκ. Για την ασφάλεια στην Ευρώπη μιλάω. Κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Στο σημείο Β. Προς μία ε, κοινή πολιτική ασφάλειας. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι μπορεί να σκεφτούμε στενότερη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής ε, ασφάλειας αλλά πριν από αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε τις δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια στα κράτη-μέλη. Μόνο λίγα κράτη-μέλη ξοδεύουν το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα. Μεταξύ άλλων είναι η Πολωνία και η Γαλλία, αλλά η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν ξοδεύουν το, ούτε καν το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα και δεν νομίζω ότι συνεισφέρουν στην ασφάλεια ολόκληρης της Υπήρου. Το ερώτημα είναι τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Γιατί αν δεν αυξήσουν τις δαπάνες τους για την ασφάλεια τα κράτη-μέλη, όλες οι άλλες διαδικασίες θα είναι εντελώς αναποτελεσματικές. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση που θα κάνει για τις δημοσιονομικές πολιτικές στα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το στοιχείο. Στις δαπάνες δηλαδή για την πολιτική άμυνα, ε, ασφάλειας. Ίσως από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Σε ό,τι αφορά τις κοινέ πολιτικές, η Μπάρμπαρα Σπινέλη. Μπάρμπαρα, ευχαριστώ. Δύο ε, προβληματισμούς επί της ουσίας και ένα ε, επί της ε, μεθοδολογίας. Μου μεγάλη εντύπωση η παρέβαση Μπροκ, που κατά την άποψή μου σωστά έδωσε έτσι μια δραματική νότα, ένα δραματικό τόνο στην κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε ότι είναι η χρονιά η αποφασιστική, που θα κρυθεί το πεπρωμένο μας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Είναι η χρονιά όπου, όπου. Εάν υπάρξει μια συνέχιση της, κατάστης της κατάστασης αδιαφάνειας, της μη ανάληψης ευθυνών, μπορεί να αποβούν πολύ επικίνδυνες. Γιατί βλέπω τι αντιλαμβάνεται ο πολίτης. Αυτό που αντιλαμβάνεται ο πολίτης αυτή είναι η πραγματικότητά του και η πραγματικότητά του μοιάζει συγκεχημένη. Και μοιάζει συγκεχημένη όχι γιατί η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομείται με βήμα όλο και πιο ταχύ. Δεν νομίζω ότι ο πολίτης ζητάει να επιβραδύνει την οικοδόμησή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ευρωπαϊκός πολίτης θέλει να καταλάβει τι συμβαίνει, να σταθεί τμήμα της οικοδόμησης αυτής. Είναι σημαντικό η έκθεση να επαναλάβει ότι αυτό που θέλουμε είναι μια πιο στενή Ευρώπη. Όλο και πιο στενή. Τώρα για να μπω σε κάτι πιο συγκεκριμένο και εγώ όπως και η ομάδα των Πρασίνων είμαι πεπισμένη ότι είναι απαραίτητο να προσφεύγουμε όλο και πιο συχνά στη ρήτρα της ε, πασαρέλας για να μπορέσουμε να περάσουμε από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία. Με αυτόν τον, πράγμα, με αυτόν τον τρόπο λαμβάνονται αποφάσεις με μεγαλύτερη διαφάνεια. Με ανησυχή ενίσχυση του ρόλου διαφόρων οργανισμών και φορέων που κατά την άποψή μου είναι χαρακτηριστική αυτής της κατάστασης αδιαφάνειας. το Eurogroup Φερρυπίν. Το οποίο δεν λογοδοτεί επαρκώς ενώπιον του Κοινοβουλίου. Δεν είναι διαφανές. Δεν έχει καν τα πρακτικά των συνεδριάσεών του. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και η αύξηση του ρόλου του με ανησυχεί για ότι αντιλαμβάνονται οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο και άλλοι οργανισμοί όπως η Frontex, που έχει νέες αρμοδιότητες σε τρίτες χώρες, αντίστοιχες με αυτές που έχει η εξωτερική πολιτική. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές για τους πρόσφυγες, ασφάλειας, τρομοκρατία, κλίμα, νομισματική ένωση, για να τα σκεφτούμε καλά όλα αυτά, σας παρακαλώ. Όχι πιεζόμενοι από τις κρίσεις. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε. Σας είμαι ευγνώμων γιατί ξοδέψατε χρόνο και θεά ουσία. Αλλά θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά καλά, για μακρόν Για τους πρόσφυγες να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν προβλήματα με τη χάρτα δικαιωμάτων με τη χάρτα για τους πρόσφυγες. Ε, το ίδιο σε ό,τι αφορά την νομισματική ένωση, την πολιτική λιτότητα. Πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα. Σε λίγο θα έχουμε και κλιματικούς πρόσφυγες. Σκεφτείτε το κι αυτό. Ίσως ε, θα ήθελα να πείτε κάτι και για αυτό το θέμα στην έκθεσή σας. Άλλο σημείο, το θέμα της μεθόδου τη μεθοδολογία σα. Η έκθεσή σας φτάνει αργά. Τη λάβαμε πολύ καθυστερημένα, δυστυχώ. Καλό θα ήταν να είχαμε το χρόνο να τη σκεφτούμε λιγάκι περισσότερο. Και να κάνουμε και μία συνάντηση με τους δύο εισηγητές, δηλαδή σκιώδεις ε, εισηγητές και βασικοί εισηγητές θα κάνουν μια συνάντηση. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση. Πώς θα ήταν χρήσιμο, μάλιστα να έχουμε περισσότερο χρόνο για τις ε, τροπολογίες, για την υποβολή τροπολογίσεων, για να μπορέσουμε να τις, ε, για να τις συζητήσουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για τη δουλειά που κάνετε και στους δύο. Πάολο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή έκθεση μπροστά μας. Δυσχερέστατο το θέμα. Δεν είναι εύκολο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις ισχύουσες συνθήκες για να βελτιώσουμε την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι το αποτέλεσμα εδώ που έχουμε μπροστά μας είναι αρκετά καλό. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ καλή δουλειά που έγινε. Και είναι ένα είδος οδικού χάρτη για μεταρρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε εντός των συνθήκων. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι έχω και εγώ τις ίδιες ανησυχίες και μοιράζομαι την απεσιοδοξία του Έλμαρ και την παρούσα κατάσταση. Οι πληροφορίες που διαθέτουμε είναι άκρος ανησυχητικές και νομίζω ότι κάποιες από τις προτινόμενες λύσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Θέλω να αναφερθώ σε δύο βασικά θέματα. Εκεί που θα επιθυμούσα μεγαλύτερη σαφήνεια. Μπορείτε να διευκρινίσετε τα εξής. Πώς βλέπετε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως βλέπω τη θέση του απλευράς θεσμικής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φαίνεται να είναι ένα σώμα, ένα ημιπροεδρικό σύστημα αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων έχουν την κατεύθυνση, δίνουν την κατεύθυνση πολιτική έχουν τη διεύθυνση στην πολιτική λοιπόν και προχωρούν πολύ μακριά όσον αφορά τις αρμοδιότητες που κανονικά έχουν στη διάθεσή τους Πώς ερμηνεύετε εσείς τη σωστή λειτουργία και την εντολή που έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει των ισχυουσών συνθήκων. Βλέπω ότι το βλέπετε με επικριτικό όμα, αλλά θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα ποια είναι η θέση σας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μετά. Θέλω να είμαι λακωνικός. Και κάτι άλλο που θα έπρεπε να τονιστεί περαιτέρω που αναφέρεται, αλλά θέλει ε, να το υπογραμμίσουμε, για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, το θέμα των μεθοριοφυλάκων και την ακτοφυλακή. Ένα είδος ε, προετοιμασίας για δυνατότητα δημιουργίας στατιωτικού δυναμικού ευρωπαϊκού ή αστυνομικού δυναμικού Έτσι θα μπορούσαμε να χτίσουμε την άμυνά μας την κοινή. Για κάποια χρόνια το σκεφτόμουν αυτό. Πάντα θεωρούσα ότι η μεθοριοφολική, με, ε, μεθοριακή, ευρωπαϊκή μεθοριοφυλακή και ακτοφυλακή ίσως δημιουργήσει τη δυνατότητα μιας κοινή άμυνας, να είναι η απαρχή μιας κοινή άμυνας. Μάλιστα μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου πρέπει να πω ότι είμαι πιο διστακτικός από ότι ήμουν θεωρούσα ότι αν και δεν ήταν άριστη πρόταση, ήταν λογική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έγινε τόσο καλά δεκτή και γι' αυτό πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε πιθανότατα πολλά προβλήματα. Αυτό ήθελα να τονίσω, το πώς ανταποκρινόμαστε στην παρούσα κρίση. Διότι η δημογραφική κρίση στο σύνολό της, η κρίση μεταναστευτική, είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, εξίσου σημαντικό στο οικονομικό. Και είναι αποφασιστική σημασία για το μέλλον της ενώσεως. Γι' αυτό πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος των θεσμών. Αυτά είχα να πω. Για την ώρα είμαι πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις μπροστά μας που υποβάλλατε. Προτάσεις πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε αν το επιθυμούμε. Αυτή την ελπίδα έχω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την παρούσα κατάσταση. Ευχαριστώ υπερβάμους Ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε, αγαπητέ εισηγητά ευχαριστώ. Δύσκολο το έργο σας μέχρι τώρα, ακόμα δυσχερέστερο το έργο σας, διότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκίνησε την πρωτοβουλία, η Επιτροπή που ξεκίνησε την πρωτοβουλία της εκθέσεως και όταν συντάσσατε την εκθέση, τα δεδομένα ήταν διαφορετικά από ό,τι τώρα, άλλαξαν σημαντικά τα δεδομένα και βλέπουμε κάποιο άγχος, κάποια ανησυχία ε, να επικρατεί στις αρχές του 2016. Αφορά τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τη δυνατότητα να αποδώσουν, deliver στα αγγλικά, να, να πετύχουν στόχους. Αυτό είναι το περιβάλλον και εκεί πρέπει να κινηθούμε και να κινηθεί η έκθεσή σας. Εγώ ανησυχώ όπως συχνά το κάνω για δύο πράγματα. Το πρώτο, με ή χωρίς αλλαγή των συνθήκων. Αν δεν μας πιάσει η μανία για την αποκατάσταση εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, ακόμα και τη ρήτρα το πασαρέλα δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε, θα αντισταθούν τα κάτι μελη Αισθανόμαστε πίεση για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Εκείνοι που γνωρίζουμε ποια είναι η σημασία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και τους κινδύνους από, από υπαναχώρηση και υποχώρηση και εγκατάλειψη στόχων διότι μαζί είμαστε ισχυρότεροι. Περισσότερα μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να πετύχουμε αποτελέσματα, οικονομικά, κοινωνικά. Και βλέπουμε ότι και η Ευρώπη δεν έχει κινητοποιηθεί αρκετά για να πετύχει αποτελέσματα. Ούτε καν στα πλαίσια των συνθήκων δεν κάνουμε αρκετά. Αυτό είναι αποφασιστική σημασίας. και επιμένω στο εξή. Η επιτυχία της COP21 θα πρέπει να μεταφραστεί σε σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Να μην θεωρήσουμε ότι μόνη απάντηση είναι το σχέδιο Juncker για την Ευρώπη. Μετά, πριν μπούμε στις λεπτομέρειες για τη λειτουργία κανενός θεσμικού οργάνου, που είναι σημαντικό για μας, που δεν είναι όμως αρκετό για να κατακτήσουμε εκ νέου τη συμφωνή γνώμη των συμπολιτών μας. Πρέπει να συναγάγουμε μαθήματα από τα γεγονότα του παρελθόντος. Φαίνεται στην προσέγγιση που ακολουθήσατε κάπως, αλλά χρειάζεται διευκρίνηση. Έχουμε την Οικονομική Νοσματική Ένωση, αλλά δεν έχουμε δώσει τα κατάλληλα εργαλεία για να επιτύχει τους στόχους της. Υπάρχει διαφορά μεταξύ φιλόδοξων στόχων και πραγματικότητα των διαθεσίμων μέσων. Και είναι θανατηφόρο αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε, ε, είμαστε, βλέπουμε μεταξύ νομισματικού και οικονομικού πυλών υπάρχει διαφορά στην Οικονομική Νομισματική Ένωση. Το ίδιο το βλέπουμε και στο Σέγγεν. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε σε μια προσέγγιση σταδιακή με μικρά βήματα. Έχουμε το Σέγγεν χωρίς να έχουμε όμως μια προσέγγιση κοινή όσον αφορά το δικαίωμα ασύλου όπως εφαρμόζεται τα κράτη-μέλη θετικής μετανάστευσης ή ελέγχου των συνόρων. Και αυτό είναι ακρογωνίως λίθος, θα έλεγα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλους τους πόρους που μας διαθέτουν συνθήκες. Όταν μπούμε τώρα στις προτάσεις, στις λεπτομέρειες, σίγουρα ανεξάρτητα από την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών θα έχετε δικαίωμα υποβληθούν πολλές τροπολογίες. Φτάνει να δει κανείς το θέμα που ξέρω κάπως Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα βλέποντας το πεδίο που πρέπει να καλύψετε. Να πάρω δύο παραδείγματα. Το δημοσιονομικό δυναμικό, οι δυνατότητες. Ο Χάιμερ Μπέργκ είναι συνεισηγητής για αυτό το θέμα και δεν ξέρουμε πώς πρέπει να προσαρμόσουμε τα πράγματα. Φαίνεται να προδικάζετε ένα πεδίο δημοσιονομικό που προκύπτει από το πλαίσιο των συνθηκών, που υπολείπεται των φιλοδοξιών που θα μπορούσαμε να έχουμε. Πρέπει να γίνει προσαρμογή. Σε σχέση με τις διάφορες επιτροπές που πρέπει να επιληφθούν των θεμάτων που αναφέρεται. Ακολουθείτε συγκεκριμένη μεθοδολογία δική σας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τέλος. Το ανέφερε ο Ελμαμπρόκ αυτό που λέω. Πώ κινητοποιούμε το 42-7, ε, το άρθρο αυτό. Διότι το 42-7, το άρθρο αυτό είναι αποτέλεσμα τη συνθήκη τη Αβώνα. Εγώ χαίρομαι που για πρώτη φορά κινητοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε το άρθρο αυτό. Το ότι δεν καταφέραμε στη συνέλευση και στις συνθήκε τη Αβώνα να το ξεπεράσουμε αυτό το όριο, ο Έλμαρ Μπροκ και εγώ ήμασταν μέλη της συνέλευσης, ξέρουμε γιατί δεν έγινε αυτό. Διότι οι συνθήκες να ξεπεράσουμε το κείμενο, τα όρια του κειμένου δεν υπήρχαν. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν, να πούμε ότι ίσως πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα αύριο, πέρα από αυτά τα όρια, αλλά να μην θεωρήσουμε ότι η προσφυγή στο άθρο αυτό αποτελούσε σφάλμα. Πρέπει να τα διαχωρίσουμε να το προσμετρήσουμε τι θα πούμε. Αντιθέτως, πολλά μπορούν να γίνουν στους συνθήκων και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα ενός πράγματος που έγινε και που αναπτύσσει τη δυνατότητα χρήσεως των συνθήκων. Θα το συζητήσουμε αυτό στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να πλαισιώσουμε σωστά πιστεύω τη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ, δεν έχω άλλους που να ζητούν το λόγο. Να δώσω το λόγο λοιπόν στους εισηγητές. Στον εισηγητή μάλλον. Ο κύριος Μπροκ, σας ευχαριστώ. Ας συγκρατήσουμε ένα πράγμα, ίσως χρειάζεται και μια αναδιατύπωση. Το λέω αυτό μετά τα όσα είπε η Περβάνς. Εμείς δεν επιθυμούμε να καθορίσουμε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Δεν είναι αυτό ο στόχος της εκθέσεως. Στόχος της εκθέσεως είναι να διαπιστώσει ποια πράγματα θα ήταν δυνατά ενδεχομένως στη βάση της συνθήκης. Εάν πολιτικά θα είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή αν θα υπάρξουν σχετικές πλειοψηφίες, τότε αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν θέλουμε σε λίγε παραγράφου να βάλουμε μέσα μια περιγραφή τη πολιτική τη Επιτροπής Προπολογισμών ή άλλων, ή άλλων επιτροπών. σω χρειάζεται να γίνει μια νέα διατύπωση για να αποφευθεί οποιαδήποτε τέτοια παρανόηση. Μιλούμε για το δυναμικό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ζήτημα πολιτική ευφυγίας ορισμένα πράγματα να μην γίνουν που ίσω να είναι δυνατά. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι δυνατόν πρέπει να γίνει κιόλα. Αυτό είναι μια παλαιά σοφία η οποία ισχύει και εδώ. Το ζήτημα αυτό της πασαρέλας που έθιξε ο κ. Γκίγκολτ και το είπε και η κυρία Σπινέτη. Πολλά από αυτά που αφορούν αποφάσεις κατά πλειοψηφία είναι ζήτημα πασαρέλ. Τα λέει και μέσα η συνθήκη. Και όμως δεν τις εκμεταλλεύει τις δυνατότητες αυτές το Συμβούλιο. Τον Σεπτέμβριο χρησιμοποιήθηκε μια δυνατότητα η οποία δινόταν ήδη εδώ και μια πενταετία από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία της συνθήκης Έρχομαι και στο θέμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου και εκεί οι υπουργοί δεν τολμούν να αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Λαμβάνουν αποφάσει μόνο εφόσον είναι δεδομένη η ομοφωνία, έτσι ώστε κανεί να μην χρειαστεί να επιστρέψει στη χώρα του ω χαμένο. Να πω το εξή όμω. Στο Συμβούλιο παραβιάζεται διαρκώ η συνθήκη τη Λισαβόνα δια τη μη χρήσεω τη δυνατότητα λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία. Και όταν δεν συμφωνούν, στο Συμβούλιο, όταν δεν χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή, δεν επιτυχάνουν συνένεση, τότε παραπέμπουν το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται πλέον να ασχοληθεί και με την τελευταία λεπτομέρεια. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όμω λαμβάνεται απόφαση πάντα μόνο με ευρωφωνία, που όμω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι νομοθετικό όργανο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισήμως δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το νομοθετικό έργο, ούτε μπορεί να εγκρίνει νομοθεσία. Πάντοτε επανέρχεται το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών, μετά καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια πρόταση και μετά να αποφασίσει το Κοινοβούλιο, ή να συναποφασίσει το Κοινοβούλιο και Πρόκειται για παραπλάνηση, πρόκειται για λεγμό παραπλάνησης. λαμβάνονται αποφάσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο και καταλήγουν τον Νοέμβριο να λάβουν αποφάσει στο Συμβούλιο Υπουργών και αν αυτό γίνει τελικά. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των ετούντων άσυλο, εδώ νομίζω δεσμεύομαστε από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την διακήρυξη της Γενέβης. Το ζήτημα, το άλλο ζήτημα είναι των προτύπων. Πώς θα αντιμετωπιστούν οι αιτούντες άσυλο. Το ίδιο για την ανταλλαγή ε, δεδομένων και πληροφοριών. Δεν λειτουργεί. Η Ευρωπόλ λαμβάνει εκθέσεις από πέντε χώρες μέλη. Και καμιά από αυτές τις πέντε χώρες μέλη δεν είναι κάποια από τις μεγάλες. Ε, και μετά διαρωτώμεθα πώς δεν λειτουργεί η αντιμετώπιση τρομοκρατίας για τον αξιότιμο Ολλανδό συνάδελφο τώρα που μακρηγόρησε. Εγώ προσωπικά δεν τον θεωρώ ακροδεξιό, ούτε απευθύνθηκα σε αυτόν. Όταν μίλησε ακροδεξιούς δεν σε αυτόν. Θεωρώ κρίμα αν ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ακροδεξιός. Εμείς δεν ζητούμε ενωμένε Πολιτείες της Ευρώπης. Ό,τι αρμοδιότητες έχουμε εδώ μας έχουν δοθεί με αποφάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι χώρες μέλη. Αρμοδιότητες μπορούν να τις δώσουν και μπορούν να τις αφαιρέσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χορηγήσει στον εαυτόν τις αρμοδιότητες. Μπορεί ωστόσο να δημιουργήσει όργανα τα οποία έχουν αρμοδιότητες, αρμοδιότητες δηλαδή που τις έχουν δοθεί από τις χώρες μέλη, αυτές να μπορούν να ασκούνται. Όταν βλέπω ότι η χώρα μου, για παράδειγμα, μέχρι τον Ιούνιο παρεμπόδιζε τις ποσοστώσεις και τώρα που χρειάζεται τις ποσοστώσεις βγαίνει και μέμφεται άλλους οι οποίοι δεν έχουν συμφωνήσει με τις ποσοστώσεις και το ίδιο ισχύει βεβαίως και για όλες τις άλλες χώρες μέλη, βλέπουμε ότι εδώ ότι ορισμένοι αρνούνται να δεχθούν κάποια νομικά εργαλεία και μετά όταν τα χρειαστούν οι ίδιοι με έμφονται τους άλλους οι δεν τα δέχονται. Το ίδιο μπορώ να συνεχίσω όπως είπα και με άλλα παραδείγματα. Ένας πόλεμος στην Μέση Ανατολή, η δυστυχία των ανθρώπων της ε, υποσαχάριας Αφρικής είναι πράγματα που δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει η Ολλανδία μόνη της. Θα χρειαστεί τη συνεργασία όλων. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να δώσετε εθνικές απαντήσεις σε θέματα όπως της αλλαγής του κλίματος, της τρομοκρατίας, της μετανάστευσης, της πείνας σε όλο τον κόσμο, των εμποδίων στο παγκόσμιο εμπόριο, αν νομίζετε ότι μία ευρωπαϊκή χώρα, μία μόνη της μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτά, να μου το πείτε τότε. Και μην ξεχνάτε την αρχή του Μονέ, ότι η κοινοτική μέθοδος είναι η βήμα-βήμα συνεργασία των χωρών η οποία οδήγησε στην νομική δεσμευτικότητα και αυτή η συνεργασία μας επέτρεψε το 2008 να αποφύγουμε την μοίρα που είχε χτυπήσει τους Ευρωπαϊκού λαού το 1929. Δεν μπορώ να απαντήσω στον Πολωνό συνάδελφο βέβαια διότι έχει αποχωρήσει να διαβάσει τα πρακτικά. Εγώ χαίρομαι πάντως που οι χώρε μέλη έχουν μια πολιτική διανομή και η Μεγάλη Βρετανία πέφτει κάτω από το 2% ενώ τις χώρες μέλη 190 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα περισσότερο από ό,τι δίνουν οι Ρώσοι ανά χρόνο και έχουμε και διπλό αριθμό στρατιωτών, δεν μιλώ για όπλα, διπλό αριθμό ε, στρατιωτών από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Με τελείως αστείο αποτέλεσμα ωστόσο, γιατί έχουμε πολύ υψηλότερο κόστος. Αν θέλουμε να κάνουμε τα λεγόμενα pooling και sharing και στους εξοπλισμούς, θα εξοικονομήσουμε πολύ περισσότερα χρήματα και με τα χρήματα που θα δαπανούμε θα μπορούμε να αποδίδουμε πολύ περισσότερα. Και με τα όσα εξοικονομήσουμε θα μπορέσουμε να σκίσουμε και κοινωνική πολιτική. Την ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο νομίζω απάντησα. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που κατά τη γνώμη μου δεν παίζει τον ρόλο του της, των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε ξεκινήσει ο ρόλος αυτός από συνεργασία τότε του Ζισκάντε με τον Χέρμουντ Σμιτ που είχαν αποφασίσει συζητώντα δίπλα στο τζάκι ότι κάπω έτσι θα πρέπει να δίνονται οι μεγάλε κατευθύνσει στην Ευρώπη και όχι να μπαίνουν και να ανακατεύονται στι τελευταίε λεπτομέρειε. Τέλο, οι συνοριακέ φρουρέ και οι ακτοφυλακέ, σωστό είναι αυτό, τα είπε όμω και η σου Μπερές αυτά και έτσι σταματώ μεν εδώ αλλά θα είχα ακόμα πάρα πάρα πολλά να πω. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις πολύ παρατηρήσεις. Θα τις λάβουμε υπόψη και σας καλώ να παρουσιάσετε και τροπολογίες. Τόσο ώστε οι ιδέες σας να απεικονιστούν και να υπάρξει μια σαφής πρόταση. Δέχομαι την ιδέα και ο Έλμαρ, ο Μπλοκ φαντάζομαι θα συμφωνεί να γίνει μια συνάντηση με τους κοιόδης συζητητές. Εξάλλου σήμερα που πολύ ε, και φαντάζομαι θα θέλουν να συζητήσουμε και ευχαριστώ όλους ως, όλους όσοι υποστήριξαν τις θετικές πτυχές της έκθεσής μας. Μερικές φορές βέβαια υπάρχουν και κάποια όρια. Ε, φτάνουμε στα όρια μας. Ε, σκέφτομαι αυτά που λέει η Περβάνος Περές. Ε, βάλαμε κάποια όρια. Δηλαδή κάποια στοιχεία τα είπαμε γενικά, όχι με λεπτομέρειες, αλλά μπορούμε να τα βελτιώσουμε αυτά τα σημεία, αν το κρίνετε απαραίτητο, αξιολογώντα και αυτά που λέτε εσεί. Ο στόχος μας ήταν να δείξουμε το εξή. Θέλω να το πω στον κύριο Χάνε μα. Όλοι μας έχουμε υπόψη ότι η συνθήκη της Λισαβόνας, όπως είπε και ο Έλμαρ, εγκρίθηκε και επικυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη, ορισμένα κράτη κάνει και δημοψηφίσματα για τη συνταγματική συνθήκη και ξανά κάναν δημοψηφίσματα για τη συνθήκη της Λισαβόνας για να την εγκρίνουν. Αποτελεί τμήμα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Όλα όσα μπορούν να γίνουν στο εσωτερικό της συνθήκης Λισαβόνας σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι ξεπερνάει τις προθέσεις διαφόρων και των πολιτών ακόμα. Είμαστε μια ένωση κρατών και όχι μια ομοσπονδία υπό την Αμερικανική έννοια ή οποιαδήποτε άλλη γενικότερη έννοια. Και οι πολίτες ενέκριναν τη Λισαβόνα μέσω των συνταγμάτων τους, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνουν τις διεθνείς συνθήκες. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζεται από τους πολίτες της αρνητικά για κάποια θέματα. Όχι γιατί δεν έχει αρκετά εργαλεία για αυτά ή γιατί δεν θέλει να τα χρησιμοποιήσει πλήρω, το οποίο είναι και αλήθεια, αλλά γιατί δεν έδωσε συγκεκριμένε και γρήγορε απαντήσει στην οικονομική κρίση. Αν μπορούσαν τα κράτη μας, μικρά, μεσαία, μεγάλα, να δώσουν ε, καταλληλότερες ε, απαντήσεις ή τα μεμονωμένα νομίσματά μας, μικρά, μεσαία και μεγάλα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση δύσκολη. Βλέπω ότι αναβιώμενες χώρες έκαναν, είναι πολύ πιο πίσω γιατί έκαναν άλλες επιλογές και πήραν έφαγα χαστούκια, ασύλτα χαστούκια από την κρίση. Είναι αλήθεια κύριε Χάνε μας ότι προχωρήσαμε πολύ στην διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και επίσης, υπάρχει και ένα θεσμικό όργανο που δεν τη δέχονται. Υπάρχουν μάλλον διάφορα θεσμικά όργανα τα οποία δεν, τα, δεν τη δέχονται όλοι. Το ίδιο ισχύει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φερρυπίν, αποφασίζει σημαντικά θέματα για τη ζωή των πολιτών ε, και όμως υπάρχουν ε, μεγάλες ε, αντιθέσεις. Το γεγονός ότι αυξάνονται οι αντιθέσεις εξαρτάται από το γεγονός ότι και η σημασία των αποφάσεων που λαμβάνουμε γίνεται όλο και πιο μεγάλη. Εγώ προέρχομαι μια χώρα που έκανε ένα δημοψήφισμα για να ψηφίσουμε την Ομοσπονδιακή Ευρώπη το 1998 το 98% των πολιτών είπε ναι. Επομένω, αισθάνομαι νομιμοποιημένη ότι πρέπει ε, να, να, να λέω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Βέβαια, ρομαντικοί ήμασταν τότε. Κανένα δεν να φανταστεί τα προβλήματα σημερινά. Τα, σημε τα πράγματα σήμερα είναι διαφορετικά. Όχι γιατί είναι σημαντικό να φτιάξουμε τα Ηνωμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γιατί πρέπει να δώσουμε κομμάτια της ε, εθνικής μα κυριαρχία και υπάρχουν δυνάμεις υπέρ και κατά. Περίπλοκη διαδικασία. Και ο κύριο Γερντόσκι, που είναι σίγουρα αντιοσκεπτικιστής και προέρχεται από ένα τέτοιο κόμμα, ε, ενώπιον όμως του θέματος της ε, κοινή άμυνα είπε ότι θα ήταν σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί καταλαβαίνει ότι η δική του χώρα δεν θα μπορούσε ποτέ από μόνη της να υπερασπιστεί τα δικά της σύνορα κοινή άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οι πολίτες δεν έχουν πρόβλημα με το γεγονός ότι υπάρχει, έχουν πρόβλημα ότι δεν υπάρχει. Αλλά θα είχαμε τη δυνατότητα να τη φτιάξουμε την κοινή άμυνα μέσω της Λισαβόνας και μας το κάναμε. Αν αύριο ασχολούμαστε, ε, μας ε, επιτίθετο κάποιος, ας μην κάνουμε υποθέσεις ποιος, αν κάποιος μας επιτίθεται, λοιπόν θα έπρεπε να ζητήσει, ε, θα έπρεπε να ζητήσουμε βοήθεια από ποιον. από τη ΣΥΠΑ. Ε, από αυτού που μπόρεσαν να φτιάξουν αυτή την ε, κοινή, το κοινό εγχείρημα ε, πριν από εμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα χρονικό. Νομίζω ότι ο κ. Κόρμπεκ όμω έχει δίκιο. ότι θα πρέπει να δώσουμε προθεσμία για τις τροπολογίες για να λάβουμε υπόψη μας και τη συζήτηση για το βρετανικό θέμα. Ε, δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Έλμαρ, αλλά μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Μπορεί να χρειαστεί να πούμε κάτι και στην εκθεσή μας για το θέμα αυτό. Ίσως μια εβδομαδούλα παραπάνω. Δεν ξέρω αν δημιουργούνται πρόβλημα με το γενικό χρονοδιάγραμμα τώρα. Αλλά εσείς, κυρία Φίμπνα, είσαστε ικανότατοι να βρείτε λύση. Έλμα, πριν πάρει το λόγο να εξηγήσω κάτι. Τι σχεδιάζουμε σήμερα. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 14 ή 15 Μαρτίου. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να συζητηθούν τροπολογίες στις 22-23 Φεβρουαρίου. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε προθεσμία υποβολή τροπολογιών την ίδια μέρα, ούτε την προηγούμενη μέρα. Το Συμβούλιο είναι 18-19, λοιπόν, τι προτείνω να κρατήσουμε τις 16 Φεβρουαρίου σε προθεσμία υποβολής τροπολογιών, αλλά να αποφασίζουμε σαν Επιτροπή ότι θα εξετάσουμε προφορικές τροπολογίες και ότι απορρεύσει ενδεχομένω από τη συμφωνία για το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου και εκεί δεν είμαστε σίγουροι τι θα γίνει. Τώρα να αναβάλουμε για ένα μήνα όταν είμαστε σίγουροι αν μέσω προφορικής τροπολογίας μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πράγματα, ίσως είναι λύση. 16 Φεβρουαρίου λοιπόν προθεσμία της τροπολογίας και 18-19 θα ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα του Συμβουλίου και τότε κάποιος προετοιμάζει προφορικές τροπολογίες στα αγγλικά και τις συμπεριλαμβάνουμε στην ψηφοφορία στις 22 και 23 Φεβρουαρίου έτσι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε όλο το πρόγραμμα για την έκθεση. Αν συμφωνείτε. Ωραία. Έλμαρ, θες να πεις κάτι. Όχι. Ναι. Μου με ενδιαφέρει το επιχείρημα ότι μπορούμε ίσως να κερδίσουμε χρόνο και να επιτρέψουμε κάποιο χρονικό περιθώριο για την περίπτωση όπου προκύψουν δυσκολίες και ενδεχομένως να σκεφτόμαστε και κάποια αναβολή. Λοιπόν, θα έλεγα να διατηρήσουμε τις προθεσμίες που είπατε, να δούμε τον Φεβρουάριο που θα έχει φτάσει η συζήτηση και αν δούμε ότι χρειαζόμαστε κάποιο περιθώριο ακόμη. Εάν μπορώ αυτό να το έχω κάπου υπόψη μου, νομίζω ότι σε ένα τέτοιο θέμα δεν θέλω να προχωρήσω με ταχείες διαδικασίες και με ενδεχόμενα ε, συμπτωματικές πλειοψηφίες. Λοιπόν, κατάμε 16 Φεβρουαρίου σε προθεσμία τροπολογιών, έτσι. Ναι, αν μάθουμε κάτι αλλάζουμε. Ναι, εντάξει, λέει ο πρόεδρος, το κάνουμε αυτό, το ώστε οι συνάδελφοι να μην καθυστερήσουν στην υποβολή τροπολογιών. Κλείνουμε με αυτό. Τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Καθυστερήσαμε κάπως δυστυχώς. Διαθεσμική συμφωνία για καλύτερη νομοθεσία. Δύο λεπτά να επενθυμίσω την ιδιαίτερη, την ειδική διαδικασία που προβλέπεται για αυτού του είδους την έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πρόταση. Στις 19 Μαΐου για τη διαθεσμική συμφωνία για καλύτερη νομοθεσία. Σαν αποτέλεσμα της αποφάσεως της διασκέψεως των Προέδρων τέλος Ιουνίου ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις. Διεξήχθησαν σε πολιτικό επίπεδο. Ο Γκίφερ Χόφστατ τις διεξήγαγε. Η διάσκεψη των Προέδρων του ανέθεσε τη θέση αυτή σε πολιτικό επίπεδο. Μετά είχαμε και τεχνική ομάδα που διοργανώθηκε από το γραφείο του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου και συνόδευσε τη διαδικασία τη διαπραγματευτική. Ασχολήθηκε με τεχνικά θέματα. Οι πρόεδροι των δύο επιτροπών της ΑΦΚΟ και της Γιούρη προσεκλήθησαν σε συναντήσεις των διασκέψεων των πρόεδρων. Ο κ. Φερχόφστατ ενημέρωνε περί των αποτελεσμάτων των επομένων ε, συναντήσεων διαπραγματεύσεων. Ο κ. Βεχόφστατ ήρθε και στην ΑΦΚΟ αναφέρθηκε στα αποτελέσματα στη, στα μισά της διαδικασίας και στις 16 Δεκεμβρίου ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Η ΑΦΚΟ έθεσε προτεραιότητες σε ένα non-paper που ενεκρίθη από τους συντονιστές και την Επιτροπή. Όταν ολοκληρώθηκαν διαπραγματεύσεις το Δεκέμβριο, η διάσκεψη των Προέδρων στις 16 Δεκεμβρίου ενέκρινε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Διάσκεψη των Προέδρων, Πρόεδρος δηλαδή του Ευρωκοινοβουλίου και επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου ενέκριναν και την, το να υπάρξουν να συνταχθούν δύο εκθέσεις όσον αφορά τη διαθεσμική αυτή συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία. Μία έκθεση επίσημη που γραμμίζεται με το εσωτερικό κανονισμό που θα υποβάλει τη διεργανική Συμφωνία στην Ολομέλεια για να δοθεί η εντολή στον πρόεδρο, η άδεια στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου να υπογράψει τη συμφωνία. Η συμφωνία ανεκρίθη από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έγινε το Δεκέμβριο. Περιμένουμε τώρα τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον στερικό κανονισμό, άρθρο 295 κυρίως, μάλλον τη συνθήκη διορθώνει πρόεδρος, σε αυτού του είδους συμφωνίες, διοργανικές συμφωνίες, όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, Το κείμενο της συμφωνίας δεν μπορεί να αλλάξει μονομερός από ένα θεσμικό όργανο. Άρα, στην περίπτωση του Ευρωκοινοβουλίου, μπορούμε μόνο να απορρίψουμε το κείμενο που είναι αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ή να το εγκρίνουμε. Αυτός είναι και ο σκοπός της εκθέσεως που συνετάχθηκε και συζητούμε σήμερα. συστήνει η έκθεση την έγκριση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων, να εγκριθούν από το Ευρωκοινοβούλιο και χορηγείται η άδεια στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου να υπογράψει τη συμφωνία. Αυτή είναι μία έκθεση. Όπως είδαμε και συζητήσαμε στους συντονιστές και όπως σας ενημέρωσα, υπάρχει επίσης η σύσταση, όπως θέλετε αποκαλέστε της διασκέψης των Προέδρων η ΑΦΚΟ ετοιμάσει άλλη έκθεση. Όπως εξήγησα το πρωί. Η έκθεση αυτή αφορά την εφαρμογή και την υλοποίηση και ερμηνεία. Όλα τα θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζητήσεων και διαπραγματεύσουν με άλλα θεσμικά όργανα να εξεταστούν τα θέματα αυτά για να, γίνει, να υπάρχει σωστή ερμηνεία από τα θεσμικά όργανα. Και το Κοινοβούλιο ίσως να χρειαστεί να αλλάξει τον εσωτερικό κανονισμό. Η δεύτερη έκθεση θα συνταχθεί τον Ρίτσαρτ Κόρμπερτ. Το δέχεται, η Γιούρι το ζητά, θα συνεργαστούμε με τη Γιούρι η οποία καλύπτει σημαντικό κομμάτι του περιεχομένου της εκθέσεως που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Αυτά για την κατάσταση. Τώρα για την έκθεση που παρουσιάζω σήμερα. Ένα τμήμα είναι το κείμενο, δύο παραρτήματα που συμμετέχουν τη Διαθεσμική Συμφωνία, το πρώτο παράρτημα και το δεύτερο κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων. Θεωρούν θεσμικά όργανα ότι η νέα διοργανική συμφωνία σέβεται την ισορροπία μεταξύ θεσμικών οργάνων και εξαρμοδιότητες και επιβεβαιώνει ότι η νέα συμφωνία γίνεται με την επιφύλαξη της συμφωνίας πλαίσιο για τη σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο ψήφισμα, στο κείμενο αυτό καθεαυτό, αναφέρονται αυτά που έχουν γίνει και υπάρχει και κατάλογος θεμάτων που απαιτούν διευκρινήσεις και δουλειά. Δεν ξέρω, είναι μακροσκελής κατάλογος, βραχής, δεν υπάρχουν κάποια πρότυπα για σύγκριση. Όμως κάποια θέματα πρέπει να τα προσέξουμε. Κυρίως όταν εξετάζουμε το θέμα της εφαρμογής και ερμηνείας της εκθέσεως. Δεν είναι αποκλειστικός ο κατάλογος όμως είναι ανοιχτός. Η διεξοδική ανάλυση θα δείξει ποια θα είναι η μορφή του καταλόγου η τελική. Στο κείμενο λοιπόν περιέχονται διάφορα σημεία τα οποία δεν μας ικανοποιούν απολύτως. Δεχόμαστε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος αλλά διατείνομαι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και το πλαίσιο εφαρμογής, να συμπεριλάβουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε κάποιες διευθετήσεις, να χρησιμοποιήσουμε τους συμπεφωνημένους μηχανισμούς με τη μέγιστη αποδοτικότητα. Αναφέρουμε τα θέματα που χρήζουν βελτιώσεων για την υλοποίηση της εκθέσεως το πλαίσιο είναι ένα από αυτά τα ζητήματα. Η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, παραδείγματι, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Τι ιδιότητε έχουν όσον αφορά τι διαπραγματεύσει. Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όμω πιστεύω, για να έχουμε σωστή ισορροπία μεταξύ νομοθετικών οργάνων. Αμοιβαία πρόσβαση στι πληροφορίε, Φερρυπίν, και στα έγγραφα στις συνεδριάσεις. Προτείνω να το εξετάσουμε το θέμα. Πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα μέσω του πλαισίου υλοποίηση και εφαρμογή. Χρειάζεται και διαφάνεια όσον αφορά το νομοθετικό έργο και τι διαδικασίες. Πώς επιτυγχάνεται αυτό. Μέσω ακριβεστέρων διατάξεων και εργαλείων που θα είναι αποτέλεσμα περαιτέρω εργασιών και βελτιώσεων όσον αφορά την αποδοτικότητα των μέτρων αυτών για να πετύχουμε διαφάνεια. Παρόμοιο σχόλιο έχω για τα εθνικά κοινοβούλια. Γενικά η στάση ήταν αρνητική των πολιτικών ομάδων όσον αφορά την αύξηση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στη διαθεσμική συμφωνία. Δεν θεωρήθηκε ότι εδώ έπρεπε να τεθεί το θέμα αυτό. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια μέσω σωστών ρυθμίσεων που θα είναι καρπός των προσπαθειών μας. Πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο και τις συνέπειες της νέας αυτής διαθεσμικής συμφωνίας, κυρίως για τον εσωτερικό κανονισμό, αλλά και τι συνέπειες υπάρχουν και για άλλες βιοργανικές διευθετήσεις που υφίστανται. Στο τέλος, Ίσως με τη βοήθεια των άλλων εισηγητών μπορούμε να προτείνουμε απλούστευση της αρχιτεκτονικής δομής των διοργανικών ρυθμίσεων που έχουμε μέχρι τώρα. Λίγο πολύ αυτού του είδους την έκθεση προτείνω να εξετάσετε. Θα ήθελα επίσης να λάβουμε υπόψη αυτά που είπε η Ολλανδική Προεδρία και η Λουξεμβουριανή Προεδρία, αυτά που ακούσαμε το πρωί και το απόγευμα, του εκπροσώπου του. πόσο εκτιμά το Συμβούλιο αυτή τη συμφωνία. Πρώτη φορά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία για ρυθμίσει μεταξύ θεσμικών οργάνων το Συμβούλιο και πόσο σημαντικό εργαλείο είναι αυτό, πόσο σοβαρό εργαλείο είναι αυτό για συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι βλέπουν αυτή τη διαθεσμική συμφωνία. Τι θα κάνουμε τώρα. Μετά τη σημερινή συζήτηση θα τεθεί προθεσμία η υποβολή τροπολογιών για αυτή την έκθεση. Όχι για την συμφωνία των αποτέλεσμα των αλλά την έκθεση της ΑΦΚΟ που ακροθυγώς παρουσίασα. Προτείνω 2 Φεβρουαρίου. 2 Φεβρουαρίου προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Και μετά συζήτηση των τροπολογιών. Λοιπόν, 2 Φεβρουαρίου προθεσμία υποβολής τροπολογιών και μετά συζήτηση των τροπολογιών 22 ή 23 Φεβρουαρίου. Ψηφοφορία όσον αφορά το σχέδιο εκθέσεως την ίδια μέρα. αν θέλετε να πάμε στην πρώτη σύνοδο του Μαρτίου. 9 με 12 του μηνός δηλαδή. Να σας υπενθυμίσω ότι όλη η διαδικασία δεν μας επιτρέπει να υποβάλουμε τροπολογίες σε σχέση με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι στην έκθεση. Που είναι όχημα η έκθεση για την αδειοδότηση του Προέδρου για να υπογράψει συμφωνία. Κάτι που απορρέει τον εσωτερικό κανονισμό και τις συνθήκες. Αυτά είναι η εισαγωγή. Ο Ρίτσαρντ απελπισμένος κουνάει το χέρι του, κάτι μας δείχνεις, ήθελες να μιλήσεις. Α, επιβεβαιώνεις ε, αυτό ότι ήσουν εσύ που αναλαμβάνεις κάτι. Ο Ρίτσαρτ. Να προσθέσω το όνομά μου στον κατάλογο των αγορητών. Αυτό είναι όλο. Είσαι ο πρώτος στον κατάλογο για να μιλήσεις. Είσαι ο πρώτος. Λοιπόν, έβαλα το όνομά μου σε μια κατάλογο μηδενικά ονόματα, με μηδέν ονόματα. Εκμόνωση των σοσιαλιστών, καλωσορίζω το κείμενο που συντάξατε ως εισηγήτρια και που παρήχθη τάχιστα. Δέχομαι το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε. Η ομάδα μου θεωρεί ότι η επιτευχής ισορροπία της συμφωνίας ήταν σημαντικότατη. Από δύο πλευρές βασικά. Χαίρομαι όλους ιδιαίτερος με τον προγραμματισμό, για τον εκ των υστέρων αξιολόγηση, όλα αυτά που αναφέρονται. Ευαίσθητο θέμα για μας ήταν η αξιολόγηση συνεπειών. Όταν θα εντάσσονται στη δικασία και πόσο πλήρης θα είναι. Χαίρομαι και χαιρόμαστε διότι τίθεται βάρος να εισάγονται αυτές οι αξιολογήσεις συνεπιών στην αρχή και όχι να υπάρχει δυνατότητα κολυσιεργίας προς το τέλος της διαδικασίας. Για να υπάρχει νέα αξιολόγηση συνεπιών θα πρέπει πρώιμα να συντάσσεται αξιολόγηση συνεπιών ξεκινώντα με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να είμαστε πλήρω ενήμεροι όσον αφορά την όλη διαδικασία που ακολουθείται. Και υπεύθυνοι οι δημοκρατικά υπεύθυνοι για τη λήψη τελική αποφάσεως να έχουν τις δέουσες πληροφορίε χωρίς εκείνοι που παράγουν την αξιολόγηση συνεπιών να έχουν το δικαίωμα αρνηση κυρία ή να μπλοκάρουν τη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί ω αποτέλεσμα. Δεύτερη πτυχή που μας ικανοποιεί και ίσως θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται πιο ξεκάθαρα στην πρόταση ψηφίσματος και θα υποβάλουμε σχετικό τροπολογία. Με άλλα λόγια, θέλω να πω το εξή. Το κόστος της μη Ευρώπης που αναφέρει η συμφωνία. Η αξιολόγηση συνεπιών δεν θα πρέπει να εξετάζει μόνο το ενδεχόμενο βάρος της νομοθεσίας για τις μικρομεσίες επιχειρήσεις και άλλους. Θα έπρεπε όμως πληρέστερα να εξετάζει το θέμα. Τι γίνεται με τον καταναλωτή, με το περιβάλλον, με τις διάφορες στοιχές της νομοθεσίας. Και ποιο είναι το κόστος της μη νομοθεσίας. Καμιά φορά βλέπετε η έλλειψη νομοθεσίας μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο διοικητικό άχθος. μιλήσμονούμε ότι όταν κάνουμε κάτι σωστό, και όχι δεν το κάνουμε πάντα σωστό, όταν το πετυχαίνουμε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορεί να περικόπτει το διοικητικό άχθος μέσω ομάδας, μιας ομάδας κανόνων για την αγορά και όχι 28 διαφορετικών ομάδων κανόνων. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο κείμενο. Συμφωνώ, συμφωνώ με αυτά που είπατε, ότι υπάρχει πράγματι ανάγκη να δοθεί συνέχεια. Αναφερθήκατε στην ξεχωριστή έκθεση που θα εξετάζει τις αναγκαίες τροπολογίες και αλλαγές που θα αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες του Κοινοβουλίου. Εγώ διατείνομαι ότι δεν είναι θέμα μόνο του εσωτερικού κανονισμού, αλλά των γενικών πρακτικών που ακολουθούμε. Ίσως το πώς λειτουργεί η διοίκησή μας και η δίευλη επικοινωνιών με τα άλλα θεσμικά όργανα. Όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν. Δεν είναι μόνο θέμα εσωτερικού κανονισμού, είναι κάτι ευρύτερο από όλα αυτά. Ε, δε μη, θα έλεγα ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα με την έκθεση και ευχαριστώ την εισηγήτρια γι' αυτό. Ράινερ Βίλεντ. Ευχαριστώ. Εγώ, αντίθετα στους προηγούμενους ομιλητές, δεν μπορώ να πω ότι εκπροσωπώ την ομάδα μου. Όμως τελευταίες μέρες το συζήτησα με κάποιους ε, συναδέλφους το θέμα αυτό και σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Ξέρω ότι τελικά είναι ή όχι πρέπει να πούμε. Αλλά σε κάποια σημεία η διατύπωση καλό θα ήταν να ήταν πιο σαφής. Υπάρχουν επίσης και κάποια πράγματα που παραλήφθηκαν εντελώς. Φερρυπίν. Διάφορα ερωτήματα που, ασκούμε, που απευθύνουν προς την Κομισιόν. Θα υποχρεώνουν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντά. Για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα ολοκληρωμένων νομικών εγγράφων. Πώς περιλαμβάνονται επίσης στην επεξεργασία τα διάφορα νομικά έγγραφα πώς εντάσσονται δηλαδή στην διαδικασία better regulation. Εγώ θα ήθελα Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβουν έστω και πολιτικά την δέσμευση να εγκύπτουν στα έγγραφα της Νομικής Επιτροπής και θα ήθελα και περισσότερη μελέτη των επιπτώσεων και ιδίω στη γραφειοκρατία και στι μικρομεσαίες επιχειρήσει πάντω γνωρίζω πώς κινούνται τα πράγματα. Δέχομαι καταρχήν ότι με την μέθοδο που προτείνει η Πρόεδρος μπορούμε δηλαδή σε βάση αυτή να εργαστούμε και να προσαρτήσουμε μια δική μας, ένα δικό μας κατάλογο ετοιμάτων. Ωστόσο, πέραν των όσων γνωρίζω, από την διαδικασία. Οφείλω να εκφράσω την έκπληξή μου για το γεγονός ότι από τη μια μεριά τα έχει πει και ο Μαυρόκ. Γνωρίζω ορισμένους που λένε ότι εδώ και εκεί χρειαζόμαστε κάποιες συμφωνίες πρώτης αναγνώσεως. Δεν γνωρίζω όμως κανέναν ευρωβουλευτή που να λέει ότι αυτή η πρακτική πρέπει να επεκταθεί. Κανένα δεν γνωρίζω. Όλοι το εξετάζουν αυτό με επιφύλαξη. βλέποντα τώρα το αρχικό κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που περιλαμβάνει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να φροντίσουμε λέει για χρήση της διαδικασίας δεύτερης αναγνωσής όταν έχει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το λέει αυτό και ενδεχομένως το δέχεται και το Συμβούλιο. Πώς θα καταφέρνουμε εμείς να αφαιρέσουμε αυτό τον πολιτικό στόχο από το έγγραφο. Δεν το κατανοώ αυτό. Και θα ήθελα να μου το εξηγήσουν αυτοί που έχουν διεξαγάγει την διαπραγμάτευση. Και δεν το κατανοώ αυτό, ειδικά σε ό,τι αφορά αυτή την πτυχή. Όταν έχουμε τόσους πολλούς φανατικούς οπαδούς της διαφάνειας. Πώς ειδικά για αυτό το θέμα στο οποίο εγκύπτουμε, μέχρι τώρα δεν μας έχει υποβληθεί κανένα έγγραφο τεσσάρων στυλών. Δεν το καταλαβαίνω. Αν είχαν, ε, αν είχαν υπάρξει άλλοι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, θα το καταλάβαινα ίσως, αλλά σε τούτη εδώ την περίπτωση το καταλαβαίνω. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω σε ορισμένα από τα θέματα που θέτεται, όσο γνωρίζω βέβαια, ε, μετά. Αλλά τώρα η κυρία Μακιντάρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν είμαι βέβαια και μέλος της Επιτροπής ΑΦΚΟ, ωστόσο έχω συμμετάσχει σε όλη την διαδικασία της επανεξέτασης του IIA εξ ονόματος της δικής μου ομάδας, της ECR, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, εξ ονόματος των οποίων και μιλώ τώρα. Πρώτον, σχόλιο για το σύνολο της διαδικασίας. Συνήθως όταν έχουμε πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή θα μεταβεί στις αρμόδιες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες καταθέτουν τροπολογίες, περνούμε από τη διαδικασία των ψηφοφοριών και φτάνουμε τελικά σε μια συνολική θέση του ε, Κοινοβουλίου και μετά προχωρούμε σε διαδικασία τριμηρούς διαλόγου, η οποία απολύει σε συμφωνία. Το ευεργέτημα της διαδικασίας των ε, επιτροπών είναι αυτή η διαφάνεια την οποία ζητούν τόσοι. Και όμως συμφωνήσαμε εμείς ως κοινοβούλιο ή πάντως στο Προεδρείο ότι αυτό θα γίνεται από ένα μόνο πρόσωπο. Και χαίρομαι που ο Γκίφερ Χόφστατ ήρθε και μίλησε στις διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες και απέσυρε ορισμένε από τις προτάσεις. Ως κοινοβούλιο να θέλουμε τώρα να υπάρχει πραγματική διαφάνεια και να έχουμε ρόλο στην διαπραγμάτευση μου φαίνεται ότι ήταν λάθος να διακολουθήσουμε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Κάτι που προέκυψε από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν με τον διαπραγματευτή και με τις πολιτικές ομάδες ήταν η ιδέα μιας ετήσιας επιθεώρησης του νομοθετικού βάρους. Και αυτό ήθελε να το δει η πολιτική ομάδα. Υπάρχουν τώρα και άλλες ιδέες χρήσιμες που θα μπορούσαν να είχαν συμπεριληφθεί και να ήταν να είχε υπάρξει μια καλύτερη αφετηρία και να είχαμε τελικά μια καλύτερη εφαρμογή της uh, Better Regulation. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει ένας αριθμός σημαντικών προτεραιοτήτων για την πολιτική μου ομάδα που δεν περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο. Πρώτα, χρειαζόμαστε ένα, μια δεσμευτική δοκιμασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την ανταγωνιστικότητα. Αυτά θέλαμε να τα δούμε. Δεσμευτική δοκιμασία για τις επιπτώσεις που θα έχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ίδιο έναν δεσμευτικό στόχο μείωσης του βάρους, των επιβαρύνσεων. Των επιβαρύνσεων του άχθους που επιβάλλουμε δια της νομοθεσίας. Πολλοί υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός στόχου μείωσης ε, του άχθους και δεν το έχουμε δει αυτό να περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Το άλλο πράγμα, ή μάλλον από τα τρία αυτά πράγματα το τρίτο, είναι η ανάγκη ενός ανεξάρτητου οργάνου, ρυθμιστικού οργάνου για την νομοθεσία. Βλέπουμε εδώ ότι σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν ότι αυτό θα είναι απόλυτο εξάρτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς θα μπορέσει να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο. Σε τρεις τομείς λοιπόν χαμένες ευκαιρίες και όπου η συμφωνία δεν πετυχαίνει τον στόχο της. Πριν τελειώσω θα ήθελα να πω ότι η ιδέα της επανεξέτασης των άλλων IIA δηλαδή των άλλων διαδεσμικών συμφωνιών αυτή με βρίσκει συμφωνία. Ε, Ευχαριστώ. Τρία σχόλια. Αν είναι σωστό αυτό που λέει ο κύριος Βίλαντ ότι βγήκε αυτή η υπόθεση των πλειώνων αναγνώσεων τότε αυτό είναι σκάνδαλο. Απαράδεκτο και αντίθετο με την δεδειγμένη βούληση της πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Και ούτε κατανοώ για ποιους λόγους. Αυτό δεν εγγυάται διαφάνεια ούτε συμμετοχή της κοινή νόμης. Να μην πέσουν τα κοινοβούλια σε αυτήν την παγίδα. Ακόμα και η Κομισιόν Εάν κάνει την πρόταση αυτή και το κοινοβούλιο δεν σπέβδει να την υιοθετήσει, ήδη βρίσκω ότι αυτό έχει μυρωδιά σκανδάλου και πρέπει να καταστεί σαφές. Για τις μικρομεσαίε επιχειρήσεις συμφωνώ με τα όσα είπε ο κ. Κόρμπετ σε ό,τι αφορά δηλαδή τις μελέτες επιπτώσεων αυτό πρέπει να γίνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα. Είναι σωστό λοιπόν εάν εξετάζονται οι οικονομικέ επιπτώσει πρέπει να εξετάζονται ειδικά και αυτέ οι οικονομικέ επιπτώσει επί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Ότι δηλαδή πάντοτε συμμετέχουν στο μεγάλο ε, πολιτικό ανοιχτό διάλογο οι μεγάλε επιχειρήσεις. όμω για τι μικρές και μεσαίε επιχειρήσεις αυτές χάνονται. Για την προστασία των συμφορών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι απόλυτα αναγκαίο να υπάρχει, να προβλεφθεί αυτή η δοκιμασία. Και αυτό δεν έχει αντίφαση με αυτό που είπε εσύ, Ρισαντ Κόρμπετ, αντιθέτως περιλαμβάνεται, ε, εμπεριέχεται και θα πρέπει να γίνει στην πράξη. Και το τρίτο είναι ένα ερώτημα που προέκυψε χθε σε συζήτηση με τον Μπεντ Λάνγκε, πρόεδρο της ΙΝΤΑ. Η είδηση είναι συμφωνίες πρέπει να διαβιβάζονται έγκαιρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι να περνούν μία περίοδο όπου θα υπνώτουν στα συρτάρια του Συμβουλίου. Αυτό ξεκαθαρίζεται στη συνθήκη. Η πρόεδρος Ιούπνερ. Κανείς άλλος δεν ζητεί το λόγο. Πολύ σύντομα, γιατί Θέλω να θέσω διάφορα θέματα. Αυτές ε, τις τροπολογίες που ανέφερε, που ανέφερε ο Ρίτσαρντ, αλλά και, τα άλλα, αυτά που είπε ο κύριος Βίλαντ και η κυρία Ματιντάια, να τα βάλουμε στο ψήφισμα ως θέματα ε, εγώ μπορώ να περιλάβω και άλλα θέματα και να τα βάλουμε στην διαπραγμάτευση με τα δύο θεσμικά όργανα στο κατάλληλο επίπεδο για να δούμε αν συμφωνούμε σε πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας. Και μπορούμε να τα περιλάβουμε με την πρόσθετη αυτή δουλειά. Και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες του αποτέλεσματος της διαπραγμάτευσης. Τώρα δεν είμαι βέβαιο ότι κατάλαβα καλά, διότι στην η πρώτη ανάγνωση είναι δικό μας προνόμιο. Εμείς αποφασίζουμε αν θα αρκεστούμε στην πρώτη ανάγνωση. Δεν λέει πουθενά τίποτα η διαθεσμική συμφωνία για το προνόμιο αυτό, το οποίο μας ανήκει, όπως είπα. Υποθέτω λοιπόν, υποθέτω ότι ίσως να μην τέθηκε το θέμα, διότι εμείς αποφασίζουμε εν τέλει. Και έτσι δεν με ενισχύει τόσο πολύ. Ασφαλώς βέβαια θα πρέπει να διεξαχθεί συζήτηση με τον Ρίτσαρτ και με τον άλλο συνάδελφο της ε, νομικής επιτροπής που ε, συμμετέχει στη συζήτηση μεταξύ ΑΦΚΟ και Γιούρι για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάντως για τα σχόλιά σας. Τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την περίπλοκη αυτή υπόθεση των ε, μελετών αντικτύπου μπαίνουν και άλλα ε, δηλαδή εδαφικές επιπτώσεις ε, και άλλα σχετικά. Αυτά όλα είναι ισοδύναμα δοκιμασιών όσον αφορά δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζονται, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ακριβώς πού, αλλά σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις, νομίζω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στην συμφωνία ως ομάδα στην οποία πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή και η οποία πρέπει να προσκαλείται στις διαβουλεύσεις για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κομισιόν. Υποθέτω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν γίνει αντικείμενο ιδιαίτερη προσοχή μέσα σε αυτή τη διαθεσμική συμφωνία. Μπορούμε ωστόσο να το βάλουμε ακόμα πιο έντονα στην έκθεση. Θα βοηθήσει πολύ επίσης εάν οι συνάδελφοί μου που έχουν ε, λίστες θεμάτων Βεβαίω δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί που δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί που αποφασίζουμε κάναμε και οι δυο ως επιτροπές ό,τι μπορούσαμε για να προωθήσουμε το θέμα και για να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στα πράγματα. Αν δεν έχετε άλλα σχόλια τώρα, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Δευτέρα Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών. Θα εξετάσουμε και θα ψηφίσουμε την έκθεση στις 22 Φεβρουαρίου. Έχουμε και το πραγματικά τελευταίο θέμα, Πασκάλ Διόν και η απαλλαγή για το 2014 για το Συμβούλιο, το Γενικό Προπολογισμό του Συμβουλίου. Πασκάλ, ορίστε γρήγορα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κατάλαβα ότι πρέπει να είμαι γρήγορο. Με δύο λόγια. Θα ξεπετάξω το θέμα. Αυτή η γνωμοδότηση, όπως ξέρετε, θέλει να περάσει μπροστά από την ε, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Ε, εδώ και 6 χρόνια έχουμε αυτό το θέμα. Το Κοινοβούλιο δεν δίνει την απαλλαγή του για τη λειτουργία του Συμβουλίου. Μιλάμε για συσσόρευση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ δημοσίου χρήματος. Είναι σημαντικό ποσό. Η γνωμοδότηση που συντάσσω είναι πολύ ρεαλιστική. Έχουμε, έτσι όπως είναι τα πράγματα, την ανικανότητα επαλήθευσης των λογαριασμών, γιατί το Συμβούλιο αρνείται απλούστατα να τους δώσει λογαριασμούς αυτούς στην Κομισιόν. Και η Κομισιόν μέσω ενός μηχανισμού που έγινε αποδεκτός άτυπα, για το πω έτσι, δίνει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να επαληθεύσει άμεσα ε, τους λογαριασμούς σε όλους τους οργανισμούς. Δεν γίνεται δηλαδή επαλήθευση σε επίπεδο κομισιόν, αλλά αφορά καμιά πενταριά θεσμικά όργανα. Η κομισιόν μας ζητάει στο Κοινοβούλιο να πάμε να επαληθεύσουμε και τους λογαριασμούς του Συμβουλίου, όμως το Συμβούλιο μας λέει «νιέτ, δεν σας δίνω αυτές τις πληροφορίες». Έχουμε δηλαδή μία καυκική κατάσταση όπου το Συμβούλιο δεν είναι στην Κομισιόν. Γιατί η Κομισιόν ζητάει από την, το Κοινοβούλιο να πάει κατευθείαν στου οργανισμού. Όταν εμεί χτυπάμε την πόρτα του Συμβουλίου, μα λέει όχι. Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, εσαί. E. Η γνωμοδότησή μου είναι νομική. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτήν την κατάσταση μη δικαίου. Επομένως, θα πρέπει να συστήσουμε να γίνει μια συζήτηση, το Συμβούλιο και η Κομισιόν να κάνουν διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί είναι παράνομη, καθαρά έναντι του ευρωπαϊκού δικαίου ε, και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των ε, δημοσίων δαπανών. Εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει, τότε, για να επανέλθω στη συζήτηση που κάναμε, τότε θα μπορούσαμε να προτείνουμε οι συνθήκε να τροποποιηθούν. Ούτω ώστε να τεθεί ένα τέρμα. Προσπάθησα να είμαι λακωνικό αλλά και περιεκτικό. And you Ζητώ συγγνώμη, ε, ζητά συγγνώμη η κυρία Τάμπαντα ε, που είναι η σκιώδη συγγήτρια, δεν μπόρεσε να είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Αλλά γενικά υποστηρίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερες πληροφορίες από το Συμβούλιο. Τώρα, αν είναι η κατάλληλη στιγμή να προτείνουμε αλλαγές συνθήκες, δεν το ξέρω. Αλλά μάλλον μπορούμε να πούμε εντάξει κάποια άλλη φορά, εν ευθέτω χρόνο θα το κάνουμε. Τέλο πάντων προσωπικά. Εμεί έχουμε αυτή την παλιά παράδοση τριών διαδικασιών και παραπάνω ε, αυτή τη ε, συμφωνία κυρίων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ότι όταν υιοθετούμε τον προπολογισμό δεν τροποποιούμε. Δεν, δεν προτείνουμε τροποποίηση στου προπολογισμού του όταν υιοθετεί το Συμβούλιο τον προπολογισμό του. Συμφωνία Ευγενική Συμφωνία Κυρίων. Πιστεύω ότι τα δύο θεσμικά όργανα θα πρέπει να ενηλικιωθούν, να πετάξουν αυτή τη Συμφωνία Κυρίων και να ελέξουν πολύ πιο σοβαρά ο ένα τον προπολογισμό του άλλου, καθώ και την απαλλαγή. Γιατί πρέπει να φοβόμαστε εμεί. Το Συμβούλιο μπορεί να σχολιάζει τι δαπάνε μα, όπω και εμεί θέλουμε να σχολιάζουμε τι δικέ του. Αλλά αυτά βεβαίω εκφράζουν τις δικές μου απόψεις και δεν εκπροσωπώ την ομάδα μου. Δεν βλέπω άλλους σκιώδεις εισηγητές, δυστυχώς, αλλά πιστεύω θα δώσουν ε, τροπολογίες. Θέλεις να σχολιάσεις αυτά που άκουσες. Όχι. 26 Ιανουαρίου, μεσημέρι, είναι η καταληκτική ημερομηνία ε, για τις τροπολογίες. Είναι περίπου δύο εβδομάδες, έτσι. Είναι μικρή έκθεση, ελπίζω να αρκεί. Μετά μπορούμε να ψηφίσουμε στις 22 Φεβρουαρίου. Αν δεν έχετε αντίρρηση. 26 Ιανουαρίου 12 η ώρα και ψηφίζουμε το Φεβρουάριο. Ευχαριστώ. Και νομίζω ότι μπορώ να κλείσω εδώ τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ.